Euh, euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας με το σημείο 25 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε τους Ούγκρους συνομιλητές μας κοντά μας και όσοι ε, είχατε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στην αποστολή στη Βουδαπέστη στα τέλη του περασμένου έτους. Θα γνωρίζετε ήδη τους υπουργούς που έχουμε σήμερα κοντά μας. Και για όλους τους άλλους όμως θα είναι μια σημαντική ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων. Θα σας κάνω εγώ μια σύντομη παρουσίαση και θα οργανώσουμε τις εργασίες μας όχι ιεραρχικά, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τη Ουγγρική κυβέρνηση, αλλά θα οργανώσουμε τις εργασίες μας βάσει των ανηλυμένων υποχρεώσεων των Υπουργών. Καταρχήν ο κύριος Μίκλο Ρέτλι, Υπουργό Εθνικών Πόρων και Κοινωνικής Πολιτικής, ο κύριος Σαντόρ Τσόμπα, Αναπληρωτής Υπουργός Απασχόλησης, που θα μας μιλήσει για θέματα πολιτικής απασχόλησης και ο κ. Ζόλταν Μπάλογ, αναπληρωτής υπουργό Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, που θα μας μιλήσει για θέματα που έχουν σχέση με τους Ρώμα. Από τις επαφές που είχαμε με την Ουγγρική Προεδρία, νομίζω ότι ο κύριος Μπαλόγ θα λάβει το λόγο πρώτος. Σας δίνω λοιπόν το λόγο αναφέροντας ε, κάτι το οποίο ίσως ήδη γνωρίζετε, ότι μόλις ψηφίσαμε την έκθεση της κυρίας Κίνκα για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Είναι μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση. Θα τη συμπεριλάβει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών στον προβληματισμό της και το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει στην Ολομέλεια μέσα στους προσεχείς μήνες. Άρα με τα θέματα τα οποία εσείς καλύπτετε βρίσκεστε στην καρδιά της επικαιρότητα για μας. Είναι το θέμα της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της μη διακριτικής μεταχείρισης, των μειονοτήτων, θέματα που μας είναι ιδιαίτερα προσφυλή. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο και σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο ομιλία για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι άλλοι υπουργοί στη συνέχεια. Πάντως θα έχετε την ευκαιρία εσείς να φύγετε πρώτος. Miniszter úr, hogy én itt ezzel a, a saját témámmal kezdhetem a mai délutáni meghallgatást. A... Ευχαριστώ, και τους άλλους υπουργούς που μου παραχώρησαν τη σειρά για να μιλήσω πρώτος. Κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας ε, θα ασχοληθούμε με τα θέματα της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της ένδυας, τη φτώχεια των παιδιών και το σύστημα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την ε, ενσωμάτωση των Ρωμά. Θα αρχίσω από το τρίτο θέμα, γιατί ε, είναι το θέμα που σήμερα θα μας απασχολήσει και δεν ε, σας αποκαλύπτω κάτι, το, ε, κάτι που είναι μυστικό αν σας πω ότι μέσα στην Ουγγρική κυβέρνηση έχουν γίνει πολλές συζητήσει σχετικά με την ενσωμάτωση των Ρωμά και για την προτεραιότητα που θα δώσουμε στο θέμα αυτό. Αποφασίσαμε ότι ναι, είναι θέμα προτεραιότητας και έχω τη χαρά σήμερα να σας μιλήσω για θέματα τα οποία επί δεκαετίες συζητούνται στην Ουγγαρία και στην κεντρική Ευρώπη γενικότερα. Εδώ και αιώνες θα έπρεπε να πούμε ότι συζητούνται τα θέματα αυτά. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν το θέμα της ενσωμάτωσης των Ρωμά στην Ευρώπη σήμερα. πολύ συχνά βλέπουμε ένα πρόβλημα χωρίς να βλέπουμε τα άτομα που συναποτελούν ε, αυτό το πρόβλημα. Αυτή η οπτική γωνία αλλάζει και πρέπει να αλλάξει στο μέλλον και θα πρέπει να θεωρούμε τους ίδιους τους Ρωμά ως συνομιλητές μας όταν προσπαθούμε να επιλύσουμε κοινά προβλήματα. Δεν είναι λοιπόν αντικείμενο του προβλήματος οι Ρωμά, είναι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτά τα οποία γίνονται. Τα προβλήματα αγγίζουν τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να εμπλέκονται και στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή προγραμμάτων που τους αφορούν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να έχουν μια παθητική στάση αλλά θα πρέπει να εμπλακούν ενεργά στην επίλυση του προβλήματος. 10 έως 12 εκατομμύρια Ρωμά ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων οι περισσότεροι θίγονται από διακριτική μεταχείριση και διαχωρισμό. Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη έχουν ληφθεί πολλές πρωτοβουλίες Και αν λάβουμε υπόψη τις συνθήκες ζωής και εργασίας των Ρωμά, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους, αντιθέτως έχει επιδεινωθεί. Είναι προκλητική ως διαπίστωση, αλλά το θέμα των Ρωμά βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη εδώ και πολλά χρόνια. Παρόλα αυτά, οι συνθήκες διαβίωσής τους έχουν επιδεινωθεί. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτείνεται μια στρατηγική πλαίσιο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρόφαση για να μην λαμβάνουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Η ενσωμάτωση των Ρωμά σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι θέμα κυρίως των κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επίσης να παρέμβουν συντονίζοντας τις εθνικές στρατηγικές. μια σημαντική απόφαση αφορά ε, τον καθορισμό του αν θα πρόκειται για απόφαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή απόφαση οικονομικών συμφερόντων. Και πρέπει να τονίσουμε ότι είναι και προς οικονομικό μας συμφέρον το να ενσωματώσουμε τους Ρωμά στην αγορά εργασίας. Η ενσωμάτωσή τους μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και να βοηθήσει να ελαφρυνθεί το βάρος των κοινωνικών συστημάτων. Η ενσωμάτωση των Ρωμά δεν αποτελεί εσωτερικό θέμα των κρατών μελών, αλλά ένα θέμα για το οποίο υπάρχει κοινό ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν γίνει πολλές ενδιαφέρουσες μελέτες επί του θέματος. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει κάνει μία μελέτη η οποία δείχνει ότι αν το ποσοστό απασχόλησης των Ρωμά έφτανε το μέσο όρο της κάθε περιφέρειας, θα είχαμε ως αποτέλεσμα αύξηση 4 6% του ΑΕΠ. Μας ενδιαφέρει λοιπόν και από οικονομική σκοπιά το να προωθήσουμε την ένταξη των Ρωμά. Υπάρχουν πολλές στρατηγικές αλλά οι στρατηγικές που μέχρι τώρα εφαρμόστηκαν δεν έδωσαν σημαντικά αποτελέσματα. Χρειάζονται μέτρα τα οποία να συνδυάζουν πολλούς τομείς, την απασχόληση, τη στέγαση, τον οικονομικό τομέα, την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης. Είναι πολύπλοκο το θέμα και χρειάζεται μια πολυσχηδή αντιμετώπιση. Ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με επιτυχία με το θέμα αυτό. Και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι την 1η Απριλίου και την 6η Απριλίου θα έχουμε τα δύο μεγάλα ραντεβού στο πλαίσιο της Προεδρίας μας για την εσωμάτωση των Ρωμά. Σε αυτές τις ημερομηνίες, 1η και 6η Απριλίου, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Λίβια Γιαρόκα, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι υπεύθυνη για την έκθεση του Κοινοβουλίου και η κυρία Κίνγκα Γκέντς από τη δική σας επιτροπή ε, έκανε την ε, συνέταξη τη γνωμοδότηση την οποία ψηφίσατε. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την έκθεση αυτή, θα μπορέσει και η έκθεση αυτή να, έχει, να επηρεάσει τις εργασίες του Συμβουλίου. Σας παρακαλώ λοιπόν και εσάς να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν, ούτω ώστε η έκθεση αυτή να εγκριθεί αν είναι δυνατόν αρχές Φεβρουαρίου και όχι το Μάρτιο. Στις 6 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλαίσιο για τις Εθνικές Στρατηγικές σχετικά με τους Ρωμά θα παρουσιαστεί και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε επί τη βάση αυτής της προτάσεως της Επιτροπής να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε τις εργασίες στο Συμβούλιο σε διάφορες ομάδες του Συμβουλίου θα συζητηθούν τα θέματα αυτά, αλλά κατά κύριο λόγο θα είναι αρμόδιο το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Και το Συμβούλιο για την Παιδεία, την Νεολαία και τον Αθλητισμό και το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης θα πρέπει να συζητήσουν το θέμα αυτό. για να διαμορφωθεί αυτή η πρόταση στρατηγικής. Στα τέλη Ιουνίου το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θα θέλαμε να είναι σε θέση να δώσει συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα μπορέσει, ελπίζουμε, να επιβεβαιώσει αυτές τις συστάσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των Ρωμά. Ποιες είναι οι δικές μας προτεραιότητες. Χρειαζόμαστε δεσμεύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών. Δεύτερον, πρέπει να προσδιορίσουμε σωστά τον πληθυσμό στόχο. Θα πρέπει να γίνει μια εξειδικευμένη στοχοθέτηση που δεν θα είναι όμως αποκλειστική. Ακόμη θα πρέπει να λυθούν υπόψη διάφορα κοινωνικά και εδαφικά θέματα. Είμαστε υπέρ της πρότασης της κυρίας Λίβια Γιαρόκα για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τις περισσότερο μειονεκτούσες μικροπεριφέρειες. Θέλουμε να μπορέσουμε ε, να συσχετίσουμε ε, την ενσωμάτωση των Ρωμά με όλες τις πολιτικές έχοντας ιδίως υπόψη τη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα διαρθρωτικά ταμεία, ούτως ώστε τα χρήματα να φτάνουν πραγματικά σε αυτούς που πρέπει να υποφεληθούν από τα κονδύλια της χρηματοδότησης. Υπάρχουν και τα άλλα θέματα που ανέφερα στην αρχή. Η φτώχεια των ε, παιδιών ε, είναι υψηλής προτεραιότητας των ε, τριών προεδριών και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που υπάρχει στον τομέα της παιδικής φτώχειας και να βελτιώσουμε τη μέθοδο ανοιχτού συντονισμού. Το 2012 θα υποβληθεί η σχετική ανακοινώση της Επιτροπής εμείς θα συγκεντρώσουμε τις εμπειρίες που υπάρχουν και θα καθορίσουμε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για το προσεχές μέλλον. Τον Ιούνιο 2011 ενδέχεται να μπορέσει το Συμβούλιο να διατυπώσει σχετικά συμπεράσματα. Η στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 μαζί με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αποτελεί μία από τις προτεραιότητες και θα το συζητήσουμε μαζί με τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε, λέει Πρόεδρος. Έχω ήδη τέσσερις ομιλητές και προς το παρόν δεν παίρνω άλλους ομιλητές στον κατάλογο. Θα κρατήσουμε τους άλλους ομιλητές για τους υπόλοιπους υπουργούς. Η κυρία Λίν, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας, ο κύριος Φάλμπρου, η κυρία Πλόμ, και η κυρία Σκιντεύσκα θα λάβουν το λόγο. Κυρία Λίν, καταρχήν. Ευχαριστώ. Μία πολύ σύντομη ερώτηση. Και ίσως ξαναπάρω το λόγο για άλλα ζητήματα με τους άλλους υπουργούς. Χαίρομαι που μιλάμε για τους Ρωμά. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια και για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά της Αναπηρίας ε, και για το ξεκίνημά της πιστεύετε ότι θα υπάρξει πρόοδο στην οριζόντια, ε, στο οριζόντιο μέτρο για την ε, ε, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Δεν υπάρχει μετάφραση στα αγγλικά. Όχι, αλλά κατάλαβα την ερώτηση, λέει ο Υπουργό. Ο κ. ¿Cuántas confederaciones... Πόσες ε, συνδικαλιστικές νομοσπονδίες υπάρχουν στην Ουγγαρία. Υφίσταται κοινωνικός διάλογος. Γιατί σε όλο το πρόγραμμα της ε, Προεδρίας δεν βλέπω καμία, ούτε μία αναφορά στον κοινωνικό διάλογο. Και τρίτη με ερώτηση είναι εξής. Είναι αλήθεια ότι στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο τροποποιούνται νόμοι με πρωτοβουλία βουλευτών προκειμένου να, αποφευχθούν, να αποφευθεί διαβούλευση με τα συνδικάτα, πιο συγκεκριμένα ο νόμος που αλλάζει τους, ε, το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο που διέπει τις απεργίες. Κυρία Πλόμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή σας. Το θέμα είναι που το Ρωμά είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα τι είπατε και για τα παιδιά. Και για τα σχέδιά σας. Ε, σύμφωνα με αυτά τα σχέδια, η στρατηγική Ρωμά ε, αγγίζει την προβληματική των ε, φτωχών παιδιών και αν ναι, τι λύση προτείνει. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για το ίδιο θέμα με την κυρία Πλόμπ, ε, το θέμα της φτώχειας, δηλαδή των παιδιών. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η Ουγγρική Προεδρία σκοπεύει να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πλήρη εκρίζωση του φαινομένου της φτώχειας των παιδιών. Θα θέλατε να απαντήσετε σε αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ. Ε, ε, λιτά όμως και σύντομα για να ακούσουμε και τους υπόλοιπους nem csak időt fogok hagyni a miniszter uraknak, hanem kérdéseket is, hiszen van néhány... Ακούστε. οι υπόλοιποι υπουργοί θα έχουν το χρόνο για να κάνουν την εισήγηση, αλλά και οι υπόλοιποι που δεν ασχολούνται με το δικό μου θέμα και για τον ε, διάλογο τον κοινωνικό και για το θέμα επίσης της στρατηγικής απέναντι στα άτομα με προβλήματα. Θα ήθελα να σας πω κάτι για το διάλογο με τα συνδικάτα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο διάλογος στα πλαίσια της για τους Ρώμα και υπάρχει συμβόλιο, συμβούλιο που οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται γιατί θεωρούμε ότι με την εργασία και με τις μελέτες, με αυτά τα δύο στοιχεία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ξεφύγουμε από το πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και το Συμβούλιο Συντονισμού Ρώμα και στο Συμβούλιο αυτό εκπροσωπούνται και τα συνδικάτα και μαζί τους προχωράμε σε αυτή τη στρατηγική εργασία για το ερώτημα της κ. Πλάμ για την φτώχεια των παιδιών και την κατάσταση των Ρώμα. Εδώ να σας δώσω στοιχεία για την Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία το ένα παιδί στα δύο είναι Ρώμα ανάμεσα στα παιδιά εκείνα που χαρακτηρίζει μια μεγάλη φτώχεια και το ποσοστό αυτό αυξάνεται. Δηλαδή όλα και περισσότερα παιδιά Ρώμα προσωπούνται. Είναι 19% και χρειάζονται ολοκληρωμένα προγράμματα για να δούμε και τα στοιχεία αυτά διάκρισης, πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν στο σχολικό σύστημα, ε, ένταξη πλήρη και κοινωνική. Όλα αυτά τα θέματα τα έχει συντάξει με ιδιαίτερη προσοχή η Προεδρία και ασχολούμεθα και με το ότι θα πρέπει από νωρίς νωρίς τα παιδιά να συμμετέχουν ε, στην όλη οργάνωση και τα παιδιά αυτά να μπορούν να προσαρμόζονται και έτσι να έχουν να αποκτούν και τα προσόντα που απαιτούνται και να μην είναι ανεργοί είναι και ειδικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν την κοινότητα των Ρώμα και πολύ συχνά ας πούμε πολύ νωρίς 12-13 χρονών τα κορίτσια των Ρώμα γίνονται μητέρες ήδη και είναι στα 35 τους γιαγιάδες και είναι δύσκολο να αποκτήσουν, να ε, καταρτιστούν, να εκπαιδευτούν, να μορφωθούν και έχουν και παιδιά ακόμα, 8 παιδιών, 8 ετών, είναι 20 ετών ο, η μητέρα και είναι 35 γιαγιά και πολλές φορές και τα τρεις αυτές γενιές είναι στη διατάξη του σχολείου. Λοιπόν, ε, και πολλές φορές εκεί δεν ασχολούνται καθόλου με τα παιδιά, το θεωρούν ε, χαμένη υπόθεση. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι πολλές φορές τα διάφορα αυτά συστήματα τα προσπαθήσαμε στην Ουγγαρία. και την υποχρεωτική εκπαίδευση επίσης. Για να παίρνουν ε, τα οικογενειακά επιδόματα θα πρέπει οπωσδήποτε να φοιτούν στο σχολείο τα παιδιά. Διαφορετικά δεν παίρνουν αυτά τα επιδόματα. Αυτό είναι έτσι ένα κίνητρο και παιδαγωγικά επίσης να μπορέσουν τα παιδιά να φοιτούν στο σχολείο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας αυτή. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Εντάξει, θα μπορούσατε να μεταβείτε και για τις υπόλοιπες ε, υποχρεώσεις και ευχαριστούμε τον Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Ελληνικής για την ε, βοήθειά του και έχει το λόγο για την παρουσίαση, την κύρια παρουσίαση, την κεντρική και το θέμα του κυρίου Ρίσα ας πούμε, στα πλαίσια αυτά θα μπορούσε να τεθεί σαν θέμα. Παρακαλούμε, μπορείτε να προχωρήσετε στην εισηγήσή σας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ μαζί με τους συναδέλφους μου προκειμένου να σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα τη Ουγγρικής Προεδρίας στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Είναι αλήθεια ότι είχα ήδη την ευκαιρία να συναντήσω ορισμένα από τα μέλη της Επιτροπής σας ε, τον περασμένο Νοέμβριο. Σήμερα θα σας μιλήσω για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είμαι πεπισμένος ότι η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι θεμελιώδου σημασία προκειμένου να καρποφορήσει η Ουγγρική Προεδρία. Ελπίζω ότι η σημερινή συνάντηση θα συνεισφέρει έτσι ώστε τους επόμενους έξι μήνες να αναζητήσουμε τις πιο κατάλληλες απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είναι πιο σημαντικό από ότι ποτέ άλλοτε να συνεργαστούμε γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση η περίοδος αυτή είναι πολύ σημαντική το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θα, έχει, θα εξετάσει την στρατηγική Ευρώπη 2020 στον τομέα της ε, απασχόλησης ε, και των κοινωνικών θεμάτων και ως Προεδρία επιθυμούμε να εστιαστούμε σε δύο πράγματα. Την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενσωμάτωση των Ρωμά. Επιπλέον, μεταξύ άλλων σημαντικών θεμάτων του ΕΠΣΚΟ, θα έχουμε ε, την ε, εφαρμογή της, ε, θα έχουμε και άλλα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής του Ευρώπη 2020, για παράδειγμα, ε, την διαχείριση του δημογραφικού ζητήματος. Επιτρέψτε μου λοιπόν τώρα να επικεντρωθώ στις προτεραιότητες μας για το τρέχον εξάμεινο. Καταρχήν να σας μιλήσω για το, τις δημογραφικές τάσεις και την συνολική διαχείριση της γύρας του πληθυσμού, την ε, εναρμόνιση της οικογενειακής ε, ζωής με την επαγγελματική ζωή. Ε, είναι θέματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και κάνουμε προσπάθειες να εξασφαλίσουμε ότι τα συνταξιδοτικά μας συστήματα θα είναι βιώσιμα. Κάτι που επίσης έχει σχέση με το, τη γύρανση του πληθυσμού. Δεν θα σας μιλήσω με πολλές λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα, διότι <clears throat> γιατί περιμένουμε ε, προτάσεις. επίσης υπάρχει και το θέμα Ευρώπη για τις οικογένειες, η οικογένεια της Ευρώπης, οι οικογένειες για την Ευρώπη και η ε, εβδομάδα των οικογενειών οι επιστήμονες, οι πολίτες και οι πολιτικοί πρέπει να ε, υποβάλουν τις ε, προτάσεις τους κατά διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Ε, θα γίνει και ένα συνέδριο εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει το θέμα της οικογένειας και της επαγγελματικής ζωής, τις νέες πολιτικές για την οικογένεια, και ιδιαίτερως πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Επίση, θα λάβει η χώρα και ένα άτυπο συνέδριο υπουργών αρμοδίων για αυτά τα θέματα. Επίσης έχουμε την δήλωση 3 συν 1, την οποία θέλουμε να υιοθετήσουμε μαζί με την Πολωνία. Το δημογραφικό, η δημογραφική πρόκληση και η απάντηση της, ε, των, των πολιτικών για την οικογένεια ε, θα βασιστούν ε, σε δουλειά προηγούμενων προεδριών αλλά και δουλειά της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία και της ε, Συμμαχίας για την Οικογένεια και τα αποτελέσματα των τριών φόρουμ, δημογραφικών φόρουμ. Η, εβδομάδα, η δημογραφική αυτή εβδομάδα θα μας επιτρέψει τον Ιούνιο να συζητήσουμε τα πορίσματά της στην ΕΠΣΚΟ, στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Η Ουγγρική Προεδρία έχει ως στόχο να υιοθετηθεί ένας αριθμός αποφάσεων σε πεδοσυμβούλιο και θα προτείνουμε μάλιστα να διοργανωθεί και ένα έτος της οικογένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Ιούνιο το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θα πάρει επίσης αποφάσεις σχετικά με την ε, δραστηριότητα γύρανση. Και θα προτείνουμε το 2014 να είναι έτος δραστηρίας γύρανσης. Είναι σημαντικό να, η δήλωση να γίνεται σε πρώτη ανάγνωση, διότι ε, οι αποφάσεις θα ληφθούν ε, από κοινού. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει. Είναι σημαντικό που ε, ο βουλευτής ε, Μαρτάν Κέσλερ ήδη ξεκίνησε τις εργασίες με την υποβολή ενός πρώτου εγγράφου. Σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα των συνταξιωτικών συστημάτων, η Ουγγρική Προεδρία θέλει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη Περιμένουμε τις πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα προκύψουν από την διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο το Μάρτιο. Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού θα προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και θα συνεισφέρουμε και εμείς την πράσινη βίβλο ενώ ταυτόχρονα θα προετοιμάσουμε και τις εργασίες που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Άλλο σημαντικό θέμα η βελτίωση της κατάστασης των αναπήρων ατόμων. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα διευκολυνόταν αν καταλαβαίναμε καλύτερα την κατάσταση αυτών των ατόμων και αν διαθέταμε συντονισμένα μέτρα υπέρ τους. Η δράση υπέρ των αναπήρων ατόμων ε, προκύπτει από την Στρατηγική Ευρώπη 2020 και είναι σημαντικό να βελτιώσουμε και να διευρύνουμε τις δυνατότητες κατάρτισης που τους δίδονται για τις δυνατότητες εκπαίδευσης και απασχόλησης. Και η κοινή γνώμη θα πρέπει να είναι και αυτή στόχος μας ε, μέσω μιας ανακοίνωσης έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να καταλάβει καλύτερα ε, τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες. Η Ουγγρική Προεδρία θα, θα διοργανώσει με τίτλο «Προκλήσεις στην πολιτική για τους ανάπηρους» ε, κατά την περίοδο 2010-2020. Θα διοργανώσω λοιπόν ένα τέτοιο ε, συνέδριο όπου θα εξετάσουμε και την συμφωνία του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αναπήρων ατόμων. Η επικύρωση αυτής της, ε, αυτού του κειμένου είναι σημαντική και γιατί πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει δικτύων ναι, θα προωθούσε μάλλον τις εξελίξεις και στην Ευρώπη. Λοιπόν, θα προωθήσουμε τα, ε, τα δικαιώματα των ε, ατόμων με αναπηρία. Δυστυχώ Δυστυχώς έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα με τη διερμηνία. On n'a plus de traduction, c'est reparti C'est bon C'est bon. Őszintén bon. hogy a magyar elnökség... Ελπίζω ότι η Ουγγρική Προεδρία θα μπορέσει να συνεργαστεί μαζί σας έτσι ώστε από κοινού να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό. θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε σε όλα τα συνέδρια τα οποία θα δωρανώσουμε για τις εκδηλώσεις. Θα σας αποστείλουμε τις προσκλήσεις εν ευθέτω χρόνο. Περιμένω τις ερωτήσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. και προτείνω να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν περισσότερο τη δική σα παρέμβαση. Προτιμάτε να ακουστούν πρώτα και οι δύο παρεμβάσει των Υπουργών για να γίνουν ερωτήσεις. Ο κ. Φάλμου. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα κηρύγματα. Έκανα τρία πολύ σαφή ερωτήματα και κανένα δεν μου απάντησε. Ρώτησα πόσε συνδικαλιστικέ συνομοσπονδίε υπάρχουν στην Ουγγαρία. Ένα. Δεύτερον, γιατί δεν αναφέρεται τίποτα για τον κοινωνικό διάλογο στο πρόγραμμα της ε, Ουγγρικής Προεδρίας και τρίτον αν ισχύει το ότι στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο αλλάζουν νόμοι, τροποποιούνται νόμοι μετά από πρωτοβουλία βουλευτών προκειμένου να αποφευχθεί η διαβούλευση με τα συνδικάτα. Δεν πήρα απάντηση. Σα είχα ξαναβάλει στον κατάλογο των ομιλητών. Μετά την παρέμβαση λοιπόν των δύο υπουργών θα είχατε την ευκαιρία να θέσετε την ερώτησή σας εκ νέου. Τώρα πάντως το άκουσαν οι Υπουργοί, άκουσαν ε, το ερώτημα που σας ενδιαφέρει. Αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό, θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Σάντορ Τσόμπα, αναπληρωτή Υπουργό Απασχόλησης, που θα μας μιλήσει για θέματα πολιτικής της απασχόλησης. Και σας παρακαλώ και εσάς να μην μακρηγορήσετε για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για το διάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίδεται και με τιμά η ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Ο Υπουργό κύριος Σαρατεγή μα ε, μίλησε για τις προκλήσει στον κοινωνικό τομέα και θα ήθελα εγώ να παρουσιάσω το πρόγραμμά μας στον τομέα της απασχόλησης. Στην τρέχουσα κοινωνική και οικονομική κατάσταση, για να μπορέσει η Ευρώπη να αποφύγει τη στασιμότητα και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στο πλαίσιο αυτό παίζει ρόλο κλειδί η πολιτική απασχόλησης, διότι είναι μια σημαντική συνιστόσα της πολιτικής της ανταγωνιστικότητας και οποιαδήποτε επένδυση σε ανθρώπινους πόρους αποτελεί απαραίτητη συνιστόσα της πολιτικής αυτής. Η πολιτική απασχόληση λοιπόν θα πρέπει να κατέχει κυρίαρχη θέση στη μακροοικονομική συζήτηση και αυτό και κατά το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η Επιτροπή σας παίζει σημαντικό ρόλο και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα αποβεί εις των κοινών μας προτεραιοτήτων. Θέλουμε να έχουμε σωστά αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης, σε στενή συνέργεια με την οικονομική διακυβέρνηση. Θα σας παρουσιάσω τώρα τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας για τον τομέα που μας ενδιαφέρει, καθώς και τα σημαντικά θέματα. Μια πρώτη προτεραιότητα για μας, ως Ουγγρική Προεδρία, είναι να επιτύχουμε στην δρομολόγηση των νέων οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να ξεκινήσουμε με επιτυχία ε, την πορεία μας προς την στρατηγική του 2020. Η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 αποτελεί ένα κοινό εργαλείο για την ενθάρρυνση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Όλοι συμφωνούμε ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής για το 2020 θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρώπη. Η απασχόληση θα ενισχυθεί μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και η ετήσια εξέταση της ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι ακριβώς θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη μαζί με απασχόληση. Θέλουμε να αποφύγουμε τους αποκλισμούς από την αγορά εργασίας. Οι στόχοι μας στο πλαίσιο της στρατηγικής για το 2020 καταγράφουν και την οδό που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχουμε τους στόχους που κοινά καθορίσαμε. Εάν η στρατηγική για το 2020 εφαρμοστεί με επιτυχία, θα μπορέσει η Ευρώπη να βγει από την κρίση και να έχει μια οικονομία βιώσιμη και πολυσυλλεκτική με υψηλή κοινωνική προστασία το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ έχει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή αυτού του πρώτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα υποβάλει σημαντικά συμπεράσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι βασικές αρχές λοιπόν θα συζητηθούν από το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ στην κοινή έκθεση για την απασχόληση και στις ε, σημαντικές συστάσεις ε, αναχώρα που επίσης θα συζητηθούν. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις ε, τροπολογίες που εσείς προσθέσατε τον, το φθινόπωρο του 2010, υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο το ε, φθινόπωρο του 2010 και θα πρέπει να υποβληθούν τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης που θα φτάσουν στην Επιτροπή μέχρι τον Απρίλιο. Και πάνω σε αυτή τη βάση θα υιοθετηθούν συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα. Οι στόχοι της Ουγγρικής Προεδρίας είναι να συνεισφέρουμε μέσω των στόχων αυτών στην επίτευξη της στρατηγικής του 2020. Η Ουγγρική Προεδρία θέλει να προωθήσει τις βασικές πρωτοβουλίες που αφορούν την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη και θα δώσουμε προτεραιότητα στις συνέργειες μεταξύ των πρωτοβουλειών και στο συμπληρωματικό τους χαρακτήρα. Η ανεργία των νέων είναι ένα λυπηρό θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη και γι' αυτό έχουμε μία εμβληματική πρωτοβουλία που ονομάζεται Youth on the Move και που δίνει πρωτοβουλία και που δίνει συγγνώμη προτεραιότητα στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Την περασμένη εβδομάδα στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό Και πραγματικά είναι κρίμα που το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών συνέπεσε με την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και έτσι δεν μπορούσε να εκπροσωπείται στη συνεδρίασή μας ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την ανεργία των νέων, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ξεπεράσει την κρίση. εφόσον δεν φαίνεται να υπάρχει αισθητή βελτίωση στη θέση των νέων στην αγορά εργασίας. Η τρέχουσα κρίση δεν θα πρέπει να διαμορφώσει το μέλλον των νέων στην αγορά εργασίας και πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε θέματα όπως η πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου, και επίσης στα άτομα που δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση. Τον Απρίλιο, επί Ουγγρικής Προεδρίας, οργανώνουμε μία διάσκεψη στην οποία θα εξετάσουμε την έξοδο από την κρίση και τη συμβολή της στην απασχόληση των νέων παράλληλα με τη στρατηγική 2020. Οι υπηρεσίε απασχόλησης των κρατών μελών θα συνεδριάσουν από τις 22 μέχρι τις 24 Ιουνίου του 2011 και στις 26 Μαΐου 2011 οργανώνουμε ένα συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θέλουμε να συζητήσουμε την συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τις προβλέψεις που γίνονται για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση οργανώνουμε ένα συνέδριο αμέσως μετά την συνάντηση των Γενικών Διευθυντών που είναι υπεύθυνοι για την επαγγελματική κατάρτιση και στο συνέδριο αυτό θα εξετάσουμε πώς μπορεί να γίνει ελκυστική για τους νέους η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και το επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τέλος, επί τη βάση των αποτελεσμάτων αυτών των δραστηριοτήτων μας, έχουμε την πρόθεση ως Ουγγρική Προεδρία να υιοθετηθούν συμπεράσματα στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του Ιουνίου Ε, και θα μας απασχολήσει το θέμα της κατάρτισης ε, και στο πλαίσιο της εκατοστής επαιτίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Το άτυπο συμβούλιο που ήδη σας ανέφερα θα συζητήσει και πάλι θέματα απασχόλησης και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα κράτη-μέλη είναι το πώς βγούμε την ε, οικονομική ανάπτυξη χωρίς αύξηση της απασχόλησης. Θέλουμε δηλαδή να διασφαλίσουμε και ανάπτυξη και παράλληλη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτές οι θέσεις απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τις απαραίτητες διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα όσον αφορά ε, τα διάφορα νομικά κείμενα, ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα για τις διάφορες προτάσεις οδηγιών. Η πρόταση οδηγίας κατά της ηλεκτρομαγνητικής ε, ακτινοβολίας για την προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ένα θέμα που επί της Προεδρίας μας θα συζητηθεί. Θα εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής το Μάρτιο και θα υποβληθεί από την Προεδρία στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ μια έκθεση πρόοδου. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τον τομέα της υγείας ιδίω για την ιονίζουσα ακτινοβολία, γνωρίζουμε ε, τι δυσκολίε και θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τι προτεραιότητε. Κατά το πρώτο εξάμεινο του 2011 θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή, σας για την, την πρότασή της για την επέκταση του πεδίου εφαρμογή έξι οδηγιών ε, που αφορά την εργασία στο πλαίσιο ε, της ναυσιπλοείας και περιμένουμε τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες ε, για την απόσπαση εργαζομένων που όμως δεν θα έχει υποβληθεί μέχρι τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2011. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2011 περιμένουμε τη δημοσίευση των οδηγιών για το χρόνο εργασίας. Επομένως θα ασχοληθεί η Πολωνική Προεδρία με το θέμα αυτό. Για την παράνομη μετανάστευση, που δεν είναι θέμα ε, του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ, υπάρχουν τρεις προτάσεις και πολλά κράτη-μέλη ζήτησαν να μην ασχοληθεί μόνο το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ, αλλά και η ομάδα εργασίας για τη μετανάστευση ε, και η Ομάδα Κοινωνικών Υποθέσεων του Συμβουλίου να ασχοληθούν επίσης με το θέμα. Όσον αφορά τις μεταφορές μεταξύ επιχειρήσεων και τους εποχιακά εργαζομένους, θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό δύο ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε. Έχω ήδη αρκετούς εγγεγραμμένους. Έχουμε μισή ωρίτσα περίπου στη διάθεσή μας. Γι' αυτό θα υποχρέωσω τον καθένα σας σε δύο λεπτά μόνο. Έτσι που είναι ήδη πέρα από το λογικό χρόνο, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά. Ε, εντάξει, θα πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα σχετικά με αυτήν την πρόεδρε όρη και σαρκάς. Köszönöm szépen a elnök asszony a szót, és meg szeretném köszönni a miniszter a ismertet. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας αυτή. Έτσι κι αλλιώς βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που εμφανίζονται στο πρόγραμμα της ε, Προεδρίας που μας απασχολούν. Θα ήθελα να τραβήξω την προσοχή σας και να πω ότι για τη στρατηγική για τα άτομα με προβλήματα ε, βλέπουμε να συντάξουμε μια έκθεση, να την παρουσιάσουμε και θα μπορούσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο ξεκινήσουμε την εργασία. Θα είχαμε την ευκαιρία δε να προχωρήσουμε και σε διαβουλεύσεις. Η κατάσταση μοιάζει όπως ε, και με αυτά που έχει να κάνει με τις νέες ε, θετικά προσόντα κλπ. Και μαζί με το Συμβούλιο μπορούμε να προωθήσουμε αυτήν την εργασία. Αρκετά αναφέρθηκαν, δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με όλα, απλά και μόνο να ζητήσω από τον κύριο Υπουργό κάποια πράγματα σχετικά με, τον, με την ενεργό γύρανση. Τι ακριβώς προβλέπετε στα προγράμματα, ποιες δραστηριότητες προβλέπετε στην ε, Ουγγρική Προεδρία και όπως το ανέφερα και στον αδελφό μου, περιμένω και την απάντησή σας, την απάντηση του κύριου Σόμπα για τα θέματα του κοινωνικού διαλόγου και πώς προβλέπει η Ουγγρική Προεδρία να προχωρήσει όσον αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για τον κύριο Τσόμπα μια ερώτηση. Με ιδιαίτερη προσοχή άκουσα το νομοθετικό του πρόγραμμα και εκ πρώτη όψεω φαίνεται ότι είναι μια οδηγία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία υπό Ουγγρική Προεδρία. Αλλά με ικανοποίηση τι άκουσα επίση, ότι θα έχουμε δύο ομάδε εργασία οι οποίε και θα ασχοληθούν ε, και θα προχωρήσουν στο δρόμο αυτό για του μετανάστες και εδώ δεν ξέρω, αλλά θα ήταν ένα βήμα ιδιαίτερα προς τα εμπρός, κύριε Τσόμπα, για αυτό το θέμα. Αν κατανοήσει το Συμβούλιο ότι αυτή η μετανάστευση δεν είναι θέμα μόνο των δικαστών και της αστυνομία, αλλά και η ένταξη των εργαζομένων. Αυτοί οι μεστανάστες εργαζόμενοι θα πρέπει να δουν αυτό το δρόμο και να δουν πώς θα ενταχθούν χωρίς φαινόμενα αποκλεισμού ή ρατσισμού. Έτσι θα λύναμε ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, στην ΕΠΣΚΟ θα πρέπει να εξεταστούν αυτά τα δύο θέματα και θα μας Πρέπει να μας υποσχεθείτε ότι τα δικαιώματα εργαζομένων μεταναστών και η ένταξη δεν θα λησμονηθούν από το Συμβούλιο και ακόμα κύριε Τσόμπα σε αυτά που είπατε εσείς να προσθέσουμε ότι είμαστε πιο προχωρημένοι σε άλλη. Αυτό το single permit και η Προεδρία θα, περάσει, θα τελειώσει η πρώτη ανάγνωση και θα πάει στο Συμβούλιο. Και η Υπουργοί Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν έλαβαν υπόψη του καθόλου το, δεν το εξέτασαν το θέμα αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα να σα παροτρύνω, αν είναι, και να έχω και τώρα μία απάντηση για αυτή την αλήψη υποχρέωση, ώστε για αυτή την ε, αποδοχή της άδεια εγκατάσταση, ότι όλα αυτά θα τα δείτε, θα τα εξετάσετε και για την κοινωνική ένταξη αυτών των εργαζομένων. Και αυτό το θέμα της μετανάστευση ε, αφορά κάθε χώρα μας και όλη την Ευρώπη, που να μην υπάρχει ε, ανταγωνισμού και κανείς ε, να μην εργάζεται χωρί κάλυψη νομική όπως αυτή που ισχύει. Αυτό είναι ζωτική σημασία για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Λίν. Και με το επόμενο. Κυρία Λίν. Ε, είχα κάνει μια ερώτηση για τα άτομα με αναπηρίες. Ε, χαίρομαι που αναφερθήκατε στην ε, σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματά τους. Όμως δεν αναφέρατε τίποτα για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, για του, τα άτομα με αναπηρίες. Ε, πώς θα μπορούσατε να μας πείτε δύο και γι' αυτό. Επίσης, να ρωτήσω το εξή Το Συμβούλιο θα απροωθήσει την οδηγία κατά των διακρίσεων και της ελεύθερης πρόσβασης υπηρεσίες και αγαθά. Υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Μετά, να σας πω το εξής. Θα ήταν ενδιαφέρον να ρωτήσω ε, για το αν θα υποστηρίξετε τη χάρτη των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων ατόμων ε, που έχουν ανάγκη φροντίδα. Επίση, για, για την οδηγία των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. Χαίρομαι που θα εξεταστεί από το Συμβούλιο. Θα θυμάστε ότι το 2004 προσπάθησα να την μπλοκάρω γιατί ε, υπήρχαν προβλήματα με, το, με τα μηχανήματα, των, ε, τα, σκάν τα scanners, ε, MRI. Ε, τώρα πια τα MRI scanners έχουν ε, εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογή, οπότε είναι καλό να προωθεί η οδηγία αυτή. Θα μπορούσατε να μας δώσετε λίγο περισσότερες πληροφορίες για το αν πιστεύετε πως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα MRI scanners στο μέλλον, αλλά τα MRI scanners ε, προωθημένης, προχωρημένης τεχνολογίας ε, θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον αυτά. Ε, παρόλο ότι τα εξαιρούμε από το πεδίο εφαρμογής. Μια διευκρίνηση λοιπόν θα ήθελα για αυτό το θέμα. Ich habe ähm, για την πολιτική απασχόληση η Ουγγρική Προεδρία έχει θέσει ω στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Νομίζω ότι η Προεδρία ε, ε, ε, του Συμβουλίου ασχολείται και με το θέμα της υψηλής φορολόγησης για τις επιχειρήσεις και νομίζω ότι έχετε πει ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλετε να έχετε μεγαλύτερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι και τους ειδικού φόρους ε, που έχετε θεσπίσει εσείς τους βλέπετε σαν μια λύση και για τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο θέμα για την ανεργία των νέων. Αναφέρατε την πρωτοβουλία Youth on the Move και είπατε τον Απρίλιο θέλετε να οργανώσετε ένα συνέδριο. Καλό είναι το ένα συνέδριο, αλλά μήπως έχετε και συγκεκριμένα μέτρα. Η Βελγική Προεδρία ήδη έλαβε κάποιες πρωτοβουλίες πολύ καλές ε, και νομίζω ότι είναι πρωτοβουλίες που προωθούν το θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι για τους δύο υπουργού έχουμε ερωτήσεις. Μήπως να μπορέσει να απαντήσει ο κύριος Τσόμπα πρώτος και μετά. Ναι, σας ευχαριστώ. Θα απαντήσω σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Πρώτα απ' όλα για τον κοινωνικό διάλογο, όπως με ρώτησαν ε, και το συνδυσμό των ε, συμφερόντων, τα συνδικάτα κλπ. Και ο κύριος Σερή αναφέρθηκε στο ίδιο θέμα και βέβαια ιδιαίτερη σημασία αποδίδομαι και σε επίπεδο κρατών μελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξαγωγή ενός πραγματικού κοινωνικού διαλόγου ε, συνεχώς και στοποθετήθηκε ακριβώς η Ουγγρική κυβέρνηση πάνω σε αυτό και στην άτυπη συνάντηση τη Δευτέρα το πρωί μπορέσαμε να συναντήσουμε τους κοινωνικούς εταίρους και ήταν ιδιαίτερα σημαντικό η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά ε, τα θέματα αυτά, τη γεννητικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και χρειάζεται συνεργασία. Καμιά κυβέρνηση από μόνη της δεν μπορεί να πετύχει. Σίγουρα θα λάβω υπόψη μου τις απόψεις ε, των κοινωνικών εταίρων. Και επίσης ε, δύο ερωτήσεις σε εθνικό επίπεδο μου τέθηκαν. Θα απαντήσω όλα μία ερώτηση για τη νέα ρύθμιση που έχει να κάνει με τις απεργίες. Το Εθνικό Συμβούλιο Διαβούλευσης όσον αφορά τα συμφέροντα και τον ΜΕ και ΔΕ είναι το ανώτατο όργανο ε, για τον κοινωνικό διάλογο και για τους μισθούς και τα υπόλοιπα θέματα αρκετά γρήγορα μπορέσαμε να, να συμφωνήσουμε. Ναι, λειτουργεί λοιπόν το σύστημα και όσον αφορά το νόμο της ρυθμίσης για την απεργία είχαμε τρεις μεταβολές που είχαν προταθεί, μία μόνο από το Εθνικό μας Κοινοβούλιο υιοθετήθηκε μετά από τις παρατηρήσεις των κοινωνικών εταίρων και απορρίφθηκαν οι υπόλοιπε δύο αλλαγέ. Μπορώ να απαντήσω και στα υπόλοιπα για τα μαγνητικά πεδία κλπ. Μπορώ να απαντήσω. Ναι, ναι, ακούστε. Ναι, ναι, αλλά αν μπορέσουμε να ακούσουμε και τις ερωτήσεις των υπολείπων μελών, μην τις χάσουμε, εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την οδηγία για την προστασία κατά των ε, μαγνητικών πεδίων, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή Θέλουμε να προχωρήσουμε, να πετύχουμε και μάλιστα σύντομα σύντομα και περιμένουμε τα έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Συμβούλιο ΕΣΚΟ. Εδώ τέθηκε ένα ερώτημα. Πότε θα κατανοήσει το Συμβούλιο το τι διακυβεύεται εκεί και τη σημασία των μεταναστών και το θέμα της κοινωνικής του ένταξης είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα αυτό. Πολύ σημαντικό για μερικά κάποια κράτη-μέλη και σίγουρα το θέμα αυτό θα παραμείνει ψηλά-ψηλά από τα πρώτα θέματα που θα εξεταθούν στην ημερήσια μας διάταξη και θα μας απασχολήσουν. Και ακόμα έχουμε και προτάσεις για τη μετανάστευση με αρκετά επιμέρους σημεία για την κοινωνική πτυχή, και συνεχώς συνεργαζόμεθα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε οι εσωτερικές πτυχές και οι κοινωνικές πτυχές όλα αυτά να ε, μπορέσουν να συνδυαστούν, να συντονιστούν. Και τώρα για την απασχόληση. Θεωρούμε ότι είναι πρωταρχικό, σημαντικότατο θέμα και δεν φτάνει να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσέξουμε και την απασχόληση. Μια οικονομική ανάπτυξη λοιπόν, αλλά εάν μειωθεί η απασχόληση ή λιμνάσει η απασχόληση, τότε δεν θα αποτελούσε λύση, γιατί ξέρουμε τι έγινε και τώρα στο πρόσφατο παρελθόν και θα το προσέξουμε. Τώρα για τους ειδικού δασμούς, ειδικού φόρους στην Η πολιτική μας απασχόλησης εντάξει μπορεί να διαφέρει βέβαια από τη μια χώρα στην άλλη και η Προεδρία η δεν θα ήθελε να προτείνει το δικό της το πρότυπο χρειάζεται να βρεθεί μια λύση για μια ε, πλήρη απασχόληση και μαζί με την οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Μου θέσατε ε, ένα ερώτημα για την στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες. Τον Ιούνιο του 2011 θέλουμε να υιοθετήσει στο Συμβούλιο συμπεράσματα ε, εν ώψη των οποίων θα διοργανώσουμε και μια διάσκεψη στην ε, Βουδαπέστη για την ε, νέα πολιτική απασχόληση 2010-2020 με τρεις άξονες την χάρτα των θεμελιδών δικαιωμάτων την Ευρωπαϊκή Στρατηγική των, και, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Ανάπηρα Άτομα πρώτον, δεύτερον απασχόληση των ανάπηρων ατόμων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και μέλλον ε, της ε, ε, Σύμβασης του ΟΗΕ. Σε ό,τι αφορά την δραστήρια γύρανση, ενεργή γύρανση, θέλουμε το 2012 να κηρυχθεί έτος ενεργούς γύρανσης θέλουμε η συμφωνία να επιτευχθεί σε πρώτη ανάγνωση έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τις προετοιμασίες πολύ γρήγορα το 2012 είναι πρώτο, πρώτον πυλών. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Θα περάσουμε σε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων, κυρία Πλόμ και μετά η κυρία Μπάουερ. Thank you very much, President. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Ρέτελη. Άκουσα την παρουσίαση σας για τις ε, πρωτοβουλίες, τη δημογραφική πρόκληση, ε, την ε, εβδομάδα υπέρ των οικογενειών κλπ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και η προώθηση της υγείας των παιδιών είναι μία από τις ναυαρχίδες ε, των προτάσεων της Ευρώπης 2020. Ε, και οι προηγούμενες προεδρίες, ε, η Ισπανία, Βέλγιο, είχαν δώσει βάρος σε αυτή την πρωτοβουλία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σχέδια έχει η Ουγγρική Προεδρία έτσι ώστε να συνεχίσει το έργο των προηγούμενων προεδριών σε αυτό το θέμα. Και να σας ρωτήσω επίσης, για ποιο λόγο πρόσφατα εισήχθη ε, η, ε, η ενιαία φορολόγηση και το οικογενειακό επίδομα το οποίο θα ωφελήσει τις οικογένειες πιο πολύ που έχουν υψηλά εισοδήματα. Οικογένειες που ήδη τα πάνε καλά οικονομικά. Ευχαριστώ. Κυρία Μπάουερ. Υπάρχει πολύ πολλά ερωτήματα. Η πάνη. το. Η Nyilvánvalóan az a, az a foglalkoztás, foglalkoztatási célkitűzés minek... Eh, Mis... Είναι προφανές ότι ο στόχος της ε, απασχόλησης... Είναι προφανές ότι ο στόχος της απασχόλησης την οποία ε, θέλουμε να φτάσουμε 75% ε, δηλαδή παντού είναι πολύ φιλόδοξος. για τις γυναίκες αυτό θα σήμαινε αύξηση απασχόληση κατά 25%. Ε, ακόμα πιο φιλόδοξο. Ε, βέβαια, η αποφάση σας είναι πολύ δικαιολογημένη. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα συμβιβάζονται οι επαγγελματικοί με την οικογενειακή ε, ζωή. Ε, θα ληφθούν υπόψη οι στόχοι της ε, Βαρκελόνης από την Ουγγρική Προεδρία. Θα γίνει η εξέταση των, των άλλων δυνατοτήτων, δηλαδή τι υπηρεσίες θα πρέπει να προσφερθούν στις οικογένειες για να πετύχουμε αυτή την αύξηση απασχόλησης. Μετά, τα βιώσιμα συνταξιδοτικά συστήματα. Ε, είναι γνωστό ότι Πήρατε αποφάσεις για τα ιδιωτικά συνταξιωτικά ταμεία. Ε, γνωρίζουμε όμως στο παρελθόν ότι έχουν υπάρξει πολλά προβλήματα με τέτοιου είδους ε, ιδιωτικές συντάξεις. Ε, πώς ε, θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συνταξιωτικών συστημάτων με αυτόν τον τρόπο. Φεντερικ Νταρντέν και μετά ο κ. Φάλμπρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, επανέρχομαι σε ένα θέμα που ήδη αναφέρθηκε και ένα, ένα σημαντικό και επίκαιρο θέμα, το θέμα των συντάξεων. Και μάλιστα εμείς βρισκόμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης της έκθεσης για την, για την Πράσινη Βίβλο και σίγουρα θα αποδώσετε ιδιαίτερη σημασία στην Πράσινη Βίβλο. Όπως είπατε, η Ουγγρική κυβέρνηση έλαβε μια σημαντική και αμφιλεγόμενη απόφαση για το δεύτερο πυλώνα της συνταξιοδότησης και μετέφερε ε, αυτές τις συνεισφορές των ε, πολιτών στον πρώτο πυλώνα. Η ερώτησή μου είναι αν η Προεδρία σας θα προτείνει και στα άλλα κράτη-μέλη μια αντίστοιχη μεταρρύθμιση και αν νομίζετε ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση μπορεί να διασφαλίσει το, τη διατήρηση του επίπεδου παροχών. Εγώ αμφιβάλλω περί αυτού. Ιδίως αν δούμε ε, το παράδειγμα της Αργεντινής, όπου διαπιστώθηκε μετά από μια τέτοια μεταρρύθμιση μείωση του επίπεδου παροχών. Ευχαριστώ. Tengo que constatar que no he recibido contestación. Ε, υπογραμμίσω ότι δεν πήρα απάντηση στις ερωτήσεις μου. Τόσο δύσκολο είναι να μου πείτε πόσες συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες υπάρχουν στην Ουγγαρία, αν υπάρχει τριμερές όργανο και αν είναι αλήθεια ότι οι νόμοι κατά των συνδικάτων εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατόπιν πρωτοβουλίας βουλευτών για να αποφευθεί ο διάλογος με τις, ε, το κοινωνικό διάλογος. Ε, είναι τόσο δύσκολο να το απαντήσετε, ακόμα και οι Τσέχοι υπουργοί θα μπορούσαν να το απαντήσουν αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και για τους στόχους της Ουγγρικής Προεδρίας που μας αναφέρατε. Ιδίως ενδιαφέρομαι για την ενεργό γύρανση. Άκουσα αυτό που είπατε ότι θέλετε ε, να προχωρήσετε για να έχουμε αποτελέσματα μέχρι το 2012 και νομίζω ότι υπάρχουν δύο θέματα και στη δική μου έκθεση και για τα οποία θα ήθελα ε, να ε, συζητήσουμε. Το θέμα του προϋπολογισμού, ποια είναι η θέση σας επ' αυτού. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αναγραφεί προϋπολογισμός στην ε, πρόταση κανονισμού της Επιτροπής και θεωρώ ότι αυτό είναι αρνητικό και νομίζω ότι και το Κοινοβούλιο γενικότερα θεωρεί αρνητικό αυτό το θέμα. Και δεύτερον, ε, όταν μιλάμε για ενεργό γύρανση, ο στόχος είναι ο τίτλος είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει να λέμε κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι εμείς ως Ευρωπαίοι, και εγώ ως νεότερος βουλευτής μπορώ να το πω αυτό, ε, για να έχουμε βιώσιμη πολιτική, η ενεργός γύρανση αρχίζει από τη στιγμή της γέννησης. Αρχίζει κανείς να γυρνάει από τη στιγμή που γεννιέται και συνεχίζεται αργότερα με τα συνταξιοδοτικά ζητήματα κλπ. Μας ενδιαφέρει η γύρανση με αξιοπρέπεια και μας ενδιαφέρει το θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών που υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει μέσα στην έκθεση. Και ένα τρίτο σημείο αυτό αποτελεί και έπαινο προς την Ουγγρική Προεδρία που αναφέρεται την πολιτική της οικογένειας ως μία από τις προτεραιότητες. Εγώ ως χριστιανοδημοκράτης το θεωρώ επίσης προτεραιότητα και χαίρομαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει όχι μόνο να μιλάμε αλλά να συνοδεύουμε τις, τα όσα λέμε και με έργα για την πολιτική που αφορά την οικογένεια και εδώ έχει σχέση η οδηγία για το χρόνο εργασίας. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα συμφιλίωσης του επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω ε, τι θα λέγατε να έχουμε μία ημέρα ελεύθερη για την οικογένεια. Και για μένα αυτή η ελεύθερη ημέρα για την οικογένεια μέσα στην εβδομάδα είναι η Κυριακή. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να το τονίσει αυτό η Ουγγρική Προεδρία. Ευχαριστώ. Θέλετε να αρχίσετε, κύριε Υπουργέ, εσείς με τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά τα θέματα της πολιτικής της οικογένειας, ε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά κρίνοντας από αυτά τα οποία ε, έχουμε ως εμπειρία στην Ουγγαρία, ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η δημογραφική πρόκληση και η οικονομική κρίση. Εξάλλου, η δημογραφική πρόκληση αποτελεί προτεραιότητα και για άλλες χώρες. Και η Σουηδία βασίστηκε στη δουλειά των προηγούμενων ε, προεδριών. Είναι σημαντικό το θέμα του ρόλου της οικογένειας. και θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες ε, να έχουν επαρκές εισόδημα μέσω της εργασίας τους. Στο πλαίσιο της οικογενειακής πολιτικής ε, παίζουν ρόλο και τα επιδόματα υπέρ των παιδιών. Χρειάζεται ένα σύστημα παρακολούθησης για κάθε μέτρο που λαμβάνεται, καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων και χρειάζεται επαρκές χρονικό διάστημα για να διαπιστώσουμε τα αποτελέσματα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι. Και θα πρέπει αντιστοίχως ε, να δούμε τα αποτελέσματα των πολιτικών μας. Για το συνταξιοδοτικό σύστημα επίσης ε, μου υποβάλλεται ερωτήσεις. η δυνατότητα παραμονής ε, στα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία ή μεταφοράς δικαιωμάτων στα δημόσια εθνικά συστήματα είναι ένα θέμα για το οποίο μέχρι τις 31 του μηνός έχουμε δώσει διορία για να μπορέσουν να αποφασίσουν οι ενδιαφερόμενοι. Και δεν θέλουμε να πάρουμε κάποια απόφαση πριν δούμε τα αποτελέσματα αυτού του μέτρου. Αυτή είναι μια λύση που δόθηκε, μια λύση που επελέγει μεταξύ άλλων για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και την πίεση στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κοινά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και πολλές ιδιαιτερότητες των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Δικός μας στόχος ε, είναι μια μεταρρύθμιση ε, του συνταξιοδοτικού συστήματος και στο μέλλον ε, θα λάβουμε και άλλα μέτρα με τελικό στόχο ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα με επαρκείς συντάξεις και με επαρκείς πόρους που θα επιτρέπουν τη χρηματοδότηση των συντάξεων για να εξασφαλίσουμε ικανοποιητική και αξιοπρεπή ε, γύρανση. Όσον αφορά την ενεργό γύρανση τώρα, θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου κάνατε. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το θέμα της χρηματοδότησης. αλλά υπάρχουν ειδικά κονδύλια για το ευρωπαϊκό έτος, για να μην χρειαστεί να προσφύγουμε σε άλλα κονδύλια και θα κάνουμε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση. Τώρα για τον τίτλο που είπατε, το πώς ε, τι τίτλο θα δώσουμε, έχετε δίκιο ότι η γύρανση αρχίζει τη στιγμή της γέννησής μας. Είμαστε ανοιχτοί για τον τίτλο που θα δοθεί στο έτος ενεργού γύρανσης αλλά δεν θα μας εμποδίσει η συζήτηση περί του τίτλου να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα μέτρα για αυτό το ειδικό έτος. Προτείνεται και μία ελεύθερη ημέρα για τις οικογένειες. Δεν το είχαμε μέσα στο πρόγραμμά μας, αλλά στην διάσκεψη που θα γίνει για την οικογένεια Ε, την εβδομάδα που προβλέπετε για το θέμα αυτό το Μάρτιο, φαντάζομαι ότι θα τεθεί και το θέμα αυτό. Όπως υπήρχαν οι προτάσεις της Βαρκελόνης, ε, ρωτήσατε αν θα υπάρξουν και προτάσεις της Βουδαπέστης. Ας περιμένουμε τα αποτελέσματα, γιατί θα έχουμε και άτυπη συνάντηση υπουργών και ίσως να προκύψει και κάτι άλλο στον τομέα αυτό. Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε τον κοινωνικό διάλογο. Δεν ε, ήθελα να βαρύνουμε την σε αυτή με εσωτερικά προβλήματα της Ουγγαρίας. Παρ' όλα αυτά να σας πω ότι το Εθνικό Συμβούλιο ε, Επίλυσης των Διαφορών είναι το το όργανο κοινωνικού διαλόγου 9 άτομα εκπροσωπούν την εργοδοσία και έξι τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τα αντιπροσωπευτικά συνδικάτα της ε, χώρας. Σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες των ε, βουλευτών, νομίζω ότι η ίδια δυνατότητα τροπολογίας νομοθεσίας ε, μέσω ε, πρωτοβουλίας βουλευτών υπάρχει σε όλα τα νομικά στήματα των κρατών ε, μελών. Ο στόχος δεν είναι να παρακάμψουμε τον κοινωνικό διάλογο, δεν είναι αυτός ο στόχος μας, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας, δεν θα μπορούσε να είναι άλλωστε. Ο κοινωνικός διάλογος είναι σημαντικός για μας όσο και για σας. Euh, κύριε Φάβρου, σας ικανοποίησε αυτή η απάντηση? Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Alors, nous, nous en venons, euh, à la... Ωραία. Εσκόμαστε στην ερώτηση για Σλοβιέσκα. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja mam pytania do... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Ρέτελη, καταρχήν. Είπατε ότι Σα ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πράσινη βίβλος για τα συνταξιωτικά ταμεία. Ερώτηση, ποια είναι η προστιθέμενη αξία του Κοινοβουλίου, τη άποψη του Κοινοβουλίου σε σχέση με την πράσινη βίβλο. Δηλαδή, ε, την άποψή μας θα την προσθέσει η Προεδρία. Επίσης, για τη Λευκή Βίβλο είπατε ότι η προτεραιότητά σας είναι οι, τα, ε, τα άτομα με αναπηρίες. Συνεπώς, δεδομένου ότι δεσμευθήκατε πως δεν θα μείνουμε στα λόγια, θα ήθελα να προετοιμάσετε κριτήρια, που θα, ε, θα ε, μέτρα που θα διευκολύνουν αυτά τα πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Κοινωνικού Ταμείου. θα δυσκολεύονται πολύ να έχουν πρόσβαση στους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ε, μην ξεχνάτε ότι ε, είναι πολύ πιο ακριβό οτιδήποτε διοργανώνουν αυτά τα άτομα, η μεταφορά, οι αίθουσες. Ε, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να έχουν πρόσβαση στα, στους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οτιδήποτε λοιπόν προτείνουν που θα τους διευκόλυνε θα ήταν πολύ καλό. Για τον Υπουργό Τσόμπα είπατε ότι θα μερινήσετε έτσι ώστε να αυξηθεί η απασχόληση των νέων. Τι έχετε προετοιμάσει, τι προβλέπετε ως καινοτόμες λύσεις. Λέω καινοτόμες έτσι στην πολιτική απασχόληση. Ενδεχομένως όχι που να απευθύνονται άμεσα στους νέους, ε, όχι μόνο στους νέους αλλά και στους ε, πιο όριμους γιατί υπάρχουν άτομα πάνω 55 ή 60 χρονών που βρίσκονται χωρίς ε, ε, δουλειά, χωρίς εργασία, ε, με όρια συνταξιοδότησης που έχουν αυξηθεί ήδη. Συνεπώς θα πρέπει και για αυτούς να προβλεφθούν μέτρα. Monsieur de Rosa, Κοφεράτη. Um, σας ευχαριστώ. Δύο σημεία. Καταρχήν ένα σημείο ενημέρωση. Άνοιξα αυτό το φυλάδιο για το πρόγραμμα τη Ουγγρική Προεδρία, Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων τη Ουγγαρία και βλέπω στο πίσω πιστόφυλλο ένα κατάλογο με χορηγού, ε, εμπορικέ εταιρείε και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πρώτη φορά βλέπω χορηγού σε φυλάδιο τη Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Audi, Volkswagen, Skoda, Saab, Citroën, Microsoft. Τι είναι αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε τι σημαίνει αυτό. Γιατί όχι, λέτε. Ναι, γιατί όχι. Το θέμα είναι ότι είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εκπροσωπούν εταιρείες ιδιωτικές. Όταν το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της Microsoft, θα επηρεαστεί η απόφασή τους από το ότι δέχτηκαν χορηγία από την εταιρεία αυτή. Ε, αυτό είναι εξωφρενικό. Και μια άλλη ερώτηση σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινή ωφελίας. Στο έγγραφο αυτό δεν αναγράφεται πουθενά το θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφελίας. Κάποιες αναφορές υπάρχουν ε, στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και ένα-δυο τέτοια σημεία. Αλλά δεδομένου ότι η Βελγική Προεδρία αφιέρωσε αρκετή δουλειά στο θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφελία ε, και διοργάνωσε και ένα συνέδριο της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπων των κρατών μελών καθώς και ευρωβουλευτών και το, συμβούλιο αυτό, το συνέδριο αυτό κατέληξε σε συστάσεις και μετά το Συμβούλιο το Δεκέμβριο κατέληξε στο ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι ουσιαστικές για να καταπολεμήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης. Μπορείτε να μας πείτε τι μέτρα θα λάβετε εσείς για να υπάρξει κάποια πρόοδος μετά τα συμπεράσματα της Βελγικής Προεδρίας επί του θέματος αυτού. Ο κύριος Κοφεράτη, η κυρία Χάρκιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για τον Υπουργό κύριο Τζόμπα να το ρωτήσω κάτι. Στην εισήγησή του πριν από λίγα λεπτά είπε ότι είναι σημαντικό, σύμφωνα με την παρατήρησή του, να εργαστεί κανείς για μια οικονομική ανάπτυξη που να πηγαίνει μαζί με την αύξηση της απασχόλησης και έτσι χρειάζεται μια ιδιαίτερη ανάπτυξη για τη χαμηλή ρυθμή ανάπτυξης όπως το γνωρίζει και εξηγεί κάθε οικονομολόγος δεν δημιουργεί επιπλέον απασχόληση και πολύ σωστά αναφέρθηκε στην ποιότητα της εργασίας όπως επίσης και στην κατάλληλη αμοιβή ανάπτυξη, νέα απασχόληση ποιοτική και βελτίωση των γενικών συνθήκων με τις οποίες διαβιούν αυτά τα άτομα. Αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος. Τώρα, μετά από όλα αυτά, πώς δικαιολογείται με την αύξηση των φόρων στις χώρες σας και μάλιστα αναδρομικά για τους δημόσιους υπαλλήλους. Τι γίνεται, μια παρόμοια επιλογή χωρίς καμία αντιστάθμιση ούτε ότι θα είναι ας πούμε σίγουροι πια για τη δουλειά τους αυτά τα άτομα. Ε, πώς θέλετε να δημιουργήσει ανάπτυξη, πώς θέλετε να παροτρύνετε αν την ε, ανάπτυξα ταυτόχρονα καταπατάτε λίγο την ε, εσωτερική κατανάλωση. κυρία Χάρκιν και μετά Γιάρικ. Χάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ουγγρική Προεδρία για την παρουσίαση που μας έκανε. Δύο ερωτήσεις. Κύριε Ρετέλη, μιλήσατε για τα άτομα με αναπηρίες και για τη συνεισφορά που μπορούν να έχουν στην κοινωνία και μιλήσατε και για βιώσιμα συνταξιοδοτικά συστήματα. Δεδομένου ότι υπάρχουν 40 άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε απασχόληση, έχετε κάποιες προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν να συνεισφέρουν προς τις βιώσιμε συντάξεις αν είχαν ε, πιο εύκολα πρόσβαση σε απασχόληση. Γιατί νομίζω ότι εδώ έχετε εν μέρη κάποια λύση στα προβλήματα. Δεύτερο σημείο, δεύτερη ερώτηση. Μία από τις προτεραιότητες που αναφέρατε είναι η μεταρρύθμιση της ε, δημοσιονομικής εποπτείας. Στον τομέα των συνταξιοδοτικών ταμείων έχετε κάποια προγράμματα, κάποια σχέδια για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής εποπτείας και εμείς έχουμε συζητήσει και το τι έχει γίνει στην Ουγγαρία με δύο, δημοσ... Ε, με δύο συνταξιδοτικά ταμεία θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη για το πώς βελτιώνεται η εποπτεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γενερίκ. Ναι, σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, προηγουμένως είπατε ότι η ανάπτυξη δεν δημιουργεί απασχόληση συμπληρωματική. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Μπορούμε να έχουμε απασχόληση με λιτή πολιτική, γιατί χρησιμοποιήσετε αυτό το η οικογένεια για την Ευρώπη και η Ευρώπη για την οικογένεια. Αυτό είπατε. Είναι νέα έννοια αυτή. Για εξηγήστε μας την και ακόμα για την ενεργό γύρανση. Τι σημαίνει αυτό, γιατί αυτόν τον όρο δεν τον καταλαβαίνω και πολύ καλά τι ακριβώς σημαίνει. Μήπως ε, να αργήσει ακόμα περισσότερο η ώρα της συνταξιοδότησης και ακόμα αληθεύει ότι στη χώρα σας ε, προτείνεται στις γυναίκες ε, που εργάζονται να επιστρέψουν στο σπίτι του τους για τρία χρόνια και υποστηρίζεται ότι θα ήταν μια καλή μέθοδος για την υπέρ της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Σρότερ και κύριε Yeah. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Προς τον κύριο Σόμπα θέλω να κάνω μια ερώτηση σε ένα σημείο που έχει σχέση με αυτά που μας ανέφερε. Και σε αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει γράφεται ότι για την οδηγία για τις αποσπάσεις θέλετε να αποφασιστεί κάποιο σύστημα στο Συμβούλιο. Έχετε καταλήξει σε συμφωνία επ' αυτού. και το σύστημα αυτό θα τροποποιήσει τις εθνικές πρακτικές στα κράτη-μέλη και τι επιπτώσεις θα υπάρχουν από αυτού. Θα μπορούσατε να μιλήσετε λίγο και για τις διαφορές απόψεων που υπάρχουν επί του θέματος. Και δεύτερον, για την παράνομη εργασία. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα ήθελα να μας πείτε ε, ποιες είναι οι προθέσεις σας επ' αυτού. Υπάρχει και η δική μου έκθεση, δεν έχουμε προχωρήσει όμως περισσότερο. Θα μπορούσατε πιο συγκεκριμένα να μας πείτε κάποια λόγια για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Köszönöm ναι, Ακούστε, δύο σύντομε ερωτήσει. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά αυτό που είπε ο κύριο Υπουργός. Συμφωνούμε νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά χρειάζεται, είναι καλύτερη πολιτική για τις συντάξει που μπορούμε να ακολουθήσουμε, να ασκήσουμε, να υπάρχει περισσότερο κόσμο στις επόμενες γιαγιές. Και ακόμα να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, αυτό που είπατε για την επιβολή φόρων και τα λοιπά στην οικογένεια, και κάνετε μια, λέτε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα παιδιά εκεί που, είναι στη μια οικογένεια με άνεση και Και, και εκείνοι που μπορούν να έχουν και ένα δικό τους διαμέρισμα, να αγοράσουν, τότε είναι πιο νόμιμη αυτή η απόκτηση παιδιών. Τι γίνεται σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Και επίσης τα οικογενειακά επιδόματα ε, είπατε ότι εξαρτώνται και τι γίνεται με τα παιδιά. Εδώ υπάρχει κάτι το αρνητικό, δηλαδή αν δεν έχουν ικανό εισόδημα, ε, τι γίνεται, μπορούν να απολαύσουν ε, μια παρόμοια με αυτή τη βοήθεια. Τι γίνεται, ποια άποψη έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, μεταρρύθμιση στις συντάξεις. Εγώ το νομίζω ότι είναι μια αντιμεταρρύθμιση. Είπατε ότι βοηθάει. Ε, νομίζω το αντίθετο. Είπατε για το δεύτερο τρίτο πυλώνα στην Ουγγαρία ότι ισχύει για να μην ε, μπαίνει στη μέση το κράτος. Και επίσης από τα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία ότι βοηθούν και αυτά στο όλο σύστημα. Και θα πρέπει κάθε σύνταξη να βασίζεται στην κοινή συνεισφορά κράτους και εργαζομένου. Τι γίνεται, πώς θα πάει όμως με τη διάρκεια ε, ισχύων αυτών, τι γίνεται για την Ουγγαρία και όλη την Ευρώπη. Κύριε Υπουργέ, εσείς είπατε ότι η οργάνωση στην ε, Στρασβούργο ήταν ε, εις βάρος διεξαγωγής των εργασιών σας και ε, σας ευχαριστούμε που το θίξατε αυτό και ότι ήταν και της Προεδρίας σας για θέματα που απασχολούν το Κοινοβούλιο είπαμε πολλά και διάφορα. Θα ήθελα να επιμείνω όμως σε δύο ειδικότερα σημεία. Το πρώτο είναι ότι το Μάιο κανονικά, δεν ξέρω πώς ακριβώς, ποια ημερομηνία, θα έχετε μια συζήτηση για το μέλος του Ταμείου Συνοχής και σημαντικό είναι η Επιτροπή αυτή να πει αυτό που έχει να πει για το μέλλον για το Μελλοντικό Κοινωνικό Ταμείο. Σας ευχαριστώ που θα το λάβετε υπόψη και να μας πείτε με ποιο τρόπο επιθυμείτε εσείς να οργανώσετε την όλη συζήτηση. Το εξάμεινο αυτό δεν θα πρόκειται για την πρώτη, το πρώτο τεστ ε, για αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και αυτό που μας έδωσε σαν κείμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας εκπλήσει σε... για πολλά πράγματα. Λέει ότι το βάρος απόδειξης ε, θα το έχουν τα κράτη με έλλειμμα. Ας αφήσουμε τώρα τι γίνεται με αυτά που έχουν πλεόνασμα που δεν ε, θα μπουν στα πλαίσια αυτής της συγκεκριμένης αλληλεγγύης, στην ανάκαμψη αυτής της συγκεκριμένης πολιτικής της οικονομικής. Αλλά καμιά φορά έχουμε την εντύπωση αυτό το βάρος απόδειξης θα βαρύνει τα θύματα της κρίσης αυτής. Οι προσανατολισμοί, οι κύριοι σε αυτές τις δέκα θέσεις προσανατολισμού που έχουν ληφθεί υπόψη, έτσι εδώ και εκεί λέει ε, περισσότερα χρόνια εργασίες χαμηλότερες συντάξεις ε, και χαμηλότερη μισθή, ξεκινώντας από αυτή τη στρατηγική που προτείνεται για την Ιρλανδία, που είναι γνωστή για την ακαμψία της αγοράς εργασίας και όλες οι περιεθνικές ε, ε, κάνω ό,τι θέλουν εκεί μέσα. Τώρα και για τι γίνεται, ότι υπό τη Βελική Προεδρία είχαμε μια πολύ σοβαρή εργασία στην Ευσκό, ώστε αυτή να μπορέσει να πει ποια είναι η αποψή τη και μέσω του βάρους που έχει στη συζήτηση αυτή τη μακροοικονομική. Εσείς ε, πώς προτίθεστε να συνεχίσετε την εργασία αυτή και αυτές οι ανησυχίες ε, που είναι των Υπουργών απασχόλησης, εργασίας απασχόλησης απέναντι στο ΕΚΟΦΗΝ και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γιατί πιστεύω, φοβάμαι ότι ουσιαστικά θα επιβεβαθούν αυτοί οι προσανατολισμοί της Επιτροπής χωρίς καμιά σημαντική αλλαγή. Τώρα δεν ξέρω ποιος από εσάς θα επιθυμούσε να λάβει πρώτος το λόγο. Κύριο Τσούμπα. Ξέρω ότι είναι πολλές ερωτήσεις που σας ετέθησαν, αλλά λίγο γρήγορα παρακαλώ απασχόληση των νέων και βελτίωση, νέες λύσεις και ενωτόμες λύσεις, ποιες δυνατότητες έχουμε. Ε, η άτυπη συνάντηση των Υπουργών είχε και αυτός θέμα στην Μεσία διάταξη. Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές, ε, τις οποίες εντοπίσαμε στα διάφορα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν. η αγορά εργασίας ε, έχει πολλά στοιχεία και εμείς στην Ουγγαρία έχουμε εντοπίσει πολλά πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ε, θέλουμε να τα μοιραστούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μόνο τους νέους, έχουμε και τους πιο όριμους ηλικιωμένους, 45, 50, 55 χρονών. Είναι αλήθεια ότι και αυτοί αποτελούν πρόκληση για μας, εξίσου μεγάλη με την απασχόληση των νέων. Θέλουμε να το δούμε και αυτό πράγματι και να βρούμε τις ε, βέλτιστες ε, πρακτικές. Πολλές ε, ερωτήσεις αφορούν την οικονομική ανάπτυξη. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Δεν είναι ερώτηση, είναι γεγονός αυτό, είναι κανόνας. Η οικονομική ανάπτυξη από ε, δεν θα βελτιώσει την κατάσταση, είναι προφανές αυτό. Ε, εσείς λέτε ότι ε, στην Ουγγαρία η φορολογία είναι πολύ ψηλή και μπορεί να δράσει ως αντικίνητρο. Οι φορολογικοί συντελεστές καθορίστηκαν αναγκαστικά σε σχετικά υψηλά επίπεδα γιατί δεν είχαμε περιθώριο ε, ελιγμών την εποχή εκείνη. Ήμασταν σε εποχή κρίσης. Όμως η φορολόγηση έτσι κι αλλιώς είναι χαμηλότερη από αυτήν άλλων κρατών μελών, πολλών άλλων κρατών μελών. Αυτό να το λάβουμε υπόψη. Σε ό,τι αφορά την ε, οδηγία της αποσπάσεις, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Άλλωστε το εξετάζει και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο εδώ και αρκετό χρόνο. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε έτσι με πολύ ε, σεβασμό αυτό το ζήτημα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου θέσατε ε, με ρωτήσατε ποια είναι η, σχέση ανάμεσα στα συνταξιωτικά ταμεία και, τους, ε, και τα άτομα με αναπηρίες. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή εργάζεται στην Λευκή, επί της Λευκής Βίβλου για την στρατηγική για τα συνταξιωτικά ταμεία και το περιεχόμενο αυτής της Λευκής Βίβλου πιθανότατα θα αλλάξει ε, ένα, θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε ένα ειδικό συνταξιωτικό ε, σύστημα για τα άτομα με αναπηρίες. Ε, είναι ένα θέμα επίμαχο στην Ευρώπη, πρέπει να σας πω. Προτείνω να περιμένουμε να δούμε την τελική μορφή της, λευκή, της πράσινης βίβλου. Σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού κοινωνική κοινής ωφελίας, Τέθηκε εδώ ένα ερώτημα. Ε, το ζήτημα αυτό δεν περιλαμβάνεται στο εγγραφό μας. Ήταν προτεραιότητα της ε, Βελγικής Προεδρίας. Δεν αποτελεί προτεραιότητα της δικής μας Προεδρίας. Γι' αυτό το λόγο κάθε χώρα έχει την ε, ευχέρεια να καθορίζει τις προτεραιότητες. ό,τι αφορά ε, το φυλάδιο αυτό δεν εκπροσωπώ το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο το τύπωσε. Νομίζω ότι ε, δε, η χορηγία δεν αφορά το ίδιο το Υπουργείο ή το κράτος, όσο ε, τη, την εκτύπωση. Ε, θα ενημερώσω το Υπουργείο Εξωτερικών για τα παραπονά σας πάντως. Σε ό,τι αφορά την καλύτερη εποπτεία των συνταξιδοτικών ταμείων, είναι αλήθεια ότι είναι απαραίτητη είναι απαραίτητη καλύτερη υποπτία όλου του χρηματοπιστωτικού τομέα και του χρηματοοικονομικού τομέα. Το κράτος δεν μπορεί να παρεμβαίνει στα συνταξιωτικά ταμεία, αλλά πρέπει να επιβάλλει την ε, εθνική νομοθεσία κάθε φορά. Μέσω της ε, εποπτείας που είναι ένα θέμα για το οποίο και το Κοινοβούλιο φαντάζομαι θα λάβει θέση πριν ε, την ε, δημοσίευση της ε, Λευκής Βίβλου από την Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά την επανειστοχή στην αγορά εργασίας ατόμων με αναπηρία, χρειάζονται θέσεις εργασίας που να είναι προσαρμοσμένες σε αυτά τα άτομα και μια κατάρτιση που να είναι προσαρμοσμένη σε αυτά τα άτομα. όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τμήμα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 γιατί για να πετύχουμε απασχόληση 75% συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να προχωρήσουμε και σε, στο θέμα της απασχόλησης των ε, ατόμων με αναπηρία. Πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, αλλά ιδιαίτερα πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης για τα άτομα με Η Ευρώπη για τις οικογένειες, οικογένειε για την Ευρώπη είναι ένα, ε, μια εκδήλωση μια εβδομάδα ε, όπου θα συζητηθεί το δημογραφικό, και το δημογραφικό πρόβλημα. Μια λύση για μας είναι να δώσουμε περισσότερη φροντίδα στις οικογένειες, να δώσουμε περισσότερη σημασία στο ρόλο και στο βάρος οικογένειας ως θεσμού. Κατά τη διάρκεια εκείνη τη εβδομάδα θα συζητήσουμε όλε αυτέ τι πτυχέ. Σε ό,τι αφορά την ενεργό γύρανση, στόχος ε, δεν είναι η αύξηση των όριων συνταξιοδότηση. Ε, ε, στόχο είναι να συζητήσουμε την πολιτική συνταξιοδότηση, <clears throat> τις πολιτικέ συνταξιοδότηση. Εσείς Είπατε ότι οι γυναίκες στην χώρα σας μπορούν να μείνουν στο σπίτι για τρία χρόνια μετά την, ε, τα τον τοκετό. Ε, εμείς το εισάγαμε αυτό από δεκαετία του 60 ε, και πράγματι οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των γεννήσεων αυτό το μέτρο. Μα ρωτάτε τι συστήνουμε στα άλλα κράτη-μέλη. Είναι δύσκολο κανεί να συστήσει οτιδήποτε σε άλλους. Ο κόσμος είναι πολύ περίπλοκος πια. Τα προβλήματα είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Κάθε χώρα θα πρέπει να εμπνευστεί από τις παραδόσεις της, την κουλτούρα της και έτσι να προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματα. Οι ουγγρικές ιδιαιτερότητες ε, ας θεωρηθούν ως απόπειρες να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να περιμένουμε και να μετρήσουμε τα αποτελέσματα αυτά. Με τα φορολογικά κίνητρα επίσης προσπαθούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των γεννήσεων. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν χρειαζόμαστε και άλλα κίνητρα για τις οικογένειες που ενδεχομένως δεν μπορούν να ε, επωφεληθούν αυτών των φοροαπαλλαγών θα πρέπει ε, να τις βοηθήσουμε και αυτές. Σε ό,τι αφορά την ε, μεταρρύθμιση των συντάξεων του συνταξιωτικού, ε, κάναμε ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε την σταθερότητα του συνταξιωτικού συστήματος. Για την βιωσιμότητα δημιουργεί πρόβλημα σε πολλά κράτη-μέλη και νομίζω θα υποβάλουμε προτάσει και για αυτό το ζήτημα κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μας. Ευχαριστώ. Κανεί από εσά όμω δεν απάντησε το ερώτημά μου. Τι θα γίνει από το ρίσκο για την προετοιμασία του Συμβουλίου της Άνοιξης από τη συμπεραίνω τίποτα δηλαδή, έτσι. Ναι. Κύριε Σούμπα. Ναι, λυπάμαι κυρία Πρόεδρε. Ναι, σημείωσα το ερώτημά σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Βελγική Προεδρία ήδη ασχολήθηκε με αυτό το θέμα ιδιαίτερα. Είχαμε πει ότι η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της ε, δεν θα δώσει όλες τις απαραίτητες λύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν την όλη μακροοικονομική συζήτηση θα θέλαμε να αποδώσουμε εκεί στο Συμβουλεύσκο να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία εταίροι μας. Ναι, θέλετε λοιπόν να συνεχίσετε ακριβώς πάνω σε αυτή τη γραμμή που χάραξε ήδη η Βελγική Προεδρία για την αξιοποίηση του ρόλου του ΕΦΣΚΟ, κυρίως απέναντι στο ΕΚΟΦΗΝ και ότι θα πρέπει να εργαστείτε γοργά για να κινητοποιήσετε τους υπουργούς όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής που έστω για ορισμένου από εμά δεν είναι μία βιώσιμη μέθοδος για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το θέμα της απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σα ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στι εργασίες μας και εύχομαι, ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάλι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Ουγγρική.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 Est-ce que je peux vous demander de quitter la salle? Παρακαλώ, μπορείτε να εξέλθετε σιωπηλά, σιωπηλά, χωρίς θόρυβο από την ε, αίθουσα. Έχουμε ήδη καθυστερήσει σχετικά με την ημερήσια μας διάταξη. Je suis totalement impuissante. Can I ask you to leave... Παρακαλώ. Μπορείτε να εξέλθετε σιωπηλά. Σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο σημείο 13 της ημερήσια μας διάταξης. Ο Στέρτζιο Κοφεράτη έχει το λόγο για τις 45 τροπολογίες για τη γνωμοδότηση για τη σημερινή κατάσταση και μελλοντικές συνέργειες για αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξης και των υπολείπων διαρθωτικών ταμείων. Το λόγο έχει ο εισηγητή μας. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ, λέει ο κύριος Κοφεράτη. Αυτές οι τροπολογίες που μας ήρθαν ε, στο κείμενο το οποίο παρουσίασα και το περι περιεχόμενό τους μας κάνουν να ελπίζουμε ότι τελικά θα καταλήξει το όλο θέμα θετικά. Δεν είναι πολλές οι τροπολογίες και ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου αυτών των τροπολογιών κατά την απόψή μου νομίζω ότι εντάσσεται, ενισχύει θετικά βέβαια όλο αυτό το σχέδιο το δικό μου. Μια παρατήρηση μόνο να κάνω και αυτό, γιατί το λέω τώρα, κάποιες δυσκολίες κάπου βλέπω εκεί στο βάθος ε, δεν έχουν σχέση με την Επιτροπή εδώ, αλλά αφορούν τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη συνέχεια στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που είναι και η, η επί της ουσίας αρμόδια Επιτροπή. Η πρότασή μου και που συμμερίζονται νομίζω όλοι ιδιαίτερα είναι ότι επιμένω στην αξία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στη χρησιμότητά του, στην αυτονομία του, στην ενίσχυσή του. Και υπάρχουν εδώ στοιχεία που είναι κατά της ενίσχυσης και είναι τα στοιχεία που μεταθέτουν την όλη προσοχή προς την εδαφική διάσταση της παρέμβασης του Ταμείου. Εντάξει, δεν είναι ότι υποτιμώ το θέμα της πρέπουσας αρμονίας εδαφικά, γεωγραφικά, μέσω της χρησιμοποίησης των Ταμείων. Αλλά κάτι να επισημάνω, ότι αρκετές φορές, πολλές φορές, τα διορθωτικό ταμεία πέρα από το κοινωνικό ταμείο χρησιμοποιήθηκαν για διαφορετικούς στόχους από ό,τι για τους στόχους για τους οποίους γεννήθηκαν και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την όλη διάκριση και να μην ε, προσφέρουμε δικαιολογίες, επιχειρήματα σε όσους επιθυμούν και εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο να μειώσουν την αξία, το βάρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έχει να κάνει με την απασχόληση και μπορεί να γίνει σημαντικότερο γιατί θα μπορούσε να ασχοληθεί και με μια νέα απασχόληση που να έχει σχέση με την αηφόρο ανάπτυξη, ορισμένες επιλογές πράσινης οικονομίας για το άμεσο μέλλον, άρα λοιπόν χώρος ανάπτυξης καινοτόμος για την απασχόληση, για την απασχόληση. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε και ότι πως ε, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα αυτό το γεωγραφικό κριτήριο. Και ίσως ε, πίσω από αυτό κρύβεται και η προσπάθεια, η κρυφή, η μη δηλωμένη, που ασκείται όμως αυτή η προσπάθεια να δυσκολέψουμε την λειτουργία και την αυτονομία του κοινωνικού ταμείου. Και τώρα είναι εδώ στην Επιτροπή που ασχολείται με την απασχόληση. Θα πρέπει να δούμε το θέμα Νομίζω ότι ε, σίγουρα απασχολεί τώρα στην απέναντι επιτροπή δεν θα ισχύει το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό χρειάζεται ακριβώ να προωθήσουμε ένα έγγραφο ιδιαίτερα αυστηρό, άκαμπτο, ας το πω έτσι, γιατί μετά στη συζήτηση που θα δεξαχθεί αλλού αυτή θα είναι διαφορετική συζήτηση από τη δική μας και όσον αφορά και τις προτάσεις και τις τροπολογίες που εδώ έχετε υποβάλει. η πρόεδρες, η κυρία Σρέτερ και μετά η κυρία Τσίμερ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοφεράτη, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς προς τα πού θέλετε να κινηθούμε. Βλέπω και τις συμβαστικές προτάσεις που τις έχουμε συζητήσει με τους σκιώτες ε, ακόμη. Ε, νομίζω ότι υπάρχει μια σαφής απόφαση του Κοινοβουλίου που λέει ότι θέλουμε να υπάρχει το κοινωνικό ταμείο κάτω από ε, το πλαίσιο όλων των διαθροτικών ταμείων, δηλαδή υπό την ίδια στέγη να είναι όλα τα διαθροτικά ταμεία και αλληλείας και γεωργίας, αλλά θέλουμε κάθε ταμείο να έχει δικούς του κανόνες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους ειδικούς στόχους που ε, ε, εκ τη γενέσεώς του έχει κάθε ταμείο. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την κοινή στέγη όλων των διαθεωτικών ταμείων. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα κοινό πλαίσιο για όλα τα ταμεία θα πρέπει να, να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε δράσεις, παραδείγματος χάρη κοινωνικού ταμείου και ταμείου για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Όταν μιλάμε για τους Ρωμά που θίγονται από συγκεκριμένα μέτρα, θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε πόρους και να συνδυάσουμε ε, τις πτυχές των διαφόρων ταμείων. Πολλές φορές έχουμε πολύ μικρά προγράμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ είναι μεγαλύτερα τα προγράμματα στο πλαίσιο άλλων διαρθρωτικών ταμείων. Βρήκαμε αυτή τη διατύπωση κατόπιν προτάσεως της ε, Προέδρου μας και νομίζω ότι είναι σημαντική η διατύπωση αυτή και θα πρέπει να παραμείνουμε στη διατύπωση αυτή. Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πόροι στο πλαίσιο των επιχειρησιακών ε, προγραμμάτων αλλά στο επίπεδο των κανονισμών θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι προσαρμοσμένα αυτά τα οποία προτείνονται για τους ε, φορείς των προγραμμάτων. Γι' αυτό σας κάνω αυτή την ερώτηση για να μας διευκρινίσετε το αν αυτά που προτείνετε συνάδουν προς τον κοινό μας στόχο η κυρία Τσίμε και ο κύριος Ντόιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό της δημογραφικής αλλαγής και της πολιτικής συνοχής. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολος τομέας και θέλουμε να βρούμε μια καινοτόμο προσέγγιση και να δώσουμε μια γνωμοδότηση από πλευράς της Επιτροπής μας. Ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα με τη γνωμοδότηση αυτή. γιατί έχουν αναπτυχθεί με τόσο διαφορετικό τρόπο οι διάφορες περιφέρειες. Γιατί σε ορισμένες περιφέρειες έχουμε περισσότερους ηλικιωμένους πάνω από το μέσο όρο σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Αυτά είναι θέματα που μπορεί να πει κανείς ότι σχετίζονται με την πολιτική για την οικογένεια και με το πώς προωθείται μια πολιτική για την οικογένεια. Αλλά κυρίως πρόκειται για διαρθρωτικές πολιτικές Θέλουμε να δούμε τι προσφέρεται στις περιφέρειες, ε, ούτως ώστε να μην φεύγουν οι νέοι, παραδείγματος χάρη, από μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Αυτά τα οποία συζητάμε είναι συνέπεια, δηλαδή φεύγουν οι νέοι φεύγουν οι νέοι με το υψηλό επίπεδο κατάρτισης από συγκεκριμένες περιφέρειες και μένουν οι πιο ηλικιωμένοι και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο τον οποίο κάποια στιγμή θέλουμε να σπάσουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια πολιτική για την οικογένεια που να λαμβάνει υπόψη της και το ποσοστό γεννητικότητας και να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση. Ένα δεύτερο σημείο και εδώ θα ήθελα ο εισηγητής ε, ε, να μου πει αν είναι θέμα ε, γλωσσικού σφάλματος, αν εγώ έχω κακή μετάφραση ή αν κάτι πρέπει να μου εξηγήσετε. Όταν μιλάμε για πολιτική για την οικογένεια, χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα για την μείωση της φτώχειας και δεν νομίζω ότι μιλάμε για το ποσοστό γεννητικότητας. Αυτό αν μπορούσατε να μου το εξηγήσετε. Δύο παρατηρήσεις λοιπόν στις οποίες θα ήθελα τη δική σας απάντηση. κύριος ε, Deutsch και μετά η κυρία Χίρς. Θέλετε το λόγο κυρία Χίρς, σας είδα καλά ή όχι. Ο κύριος Deutsch. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Κοφεράτη προετοίμασε αυτή την έκθεση την οποία χαιρετίζω ως της του ΕΛΚ. Ε, διαβάντας τις ε, προτάσεις τροπολογίας που είχε υποβάλει, ε, προ... μου δημιουργήθηκαν κάποιες μικρές απορίες και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να τις διευκρινίσουμε σήμερα. Κατά τη διάρκεια τη εισαγωγή του κ. Κοφεράτη, αυτέ οι απορίε, αυτά τα ερωτηματικά είναι πιο ισχυρά. Πιστεύω ότι είναι λάθος, θα ήταν λάθος να αμφισβητήσουμε πράγματα ε, βάζοντας ένα ερωτηματικό στο τέλος μιας φράσης. Α βάλουμε μια τελεία, α βάλουμε ένα θαυμαστικό, αλλά όχι ερωτηματικό, σε ό,τι αφορά το μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, θα έχει, έχει και έχει ήδη συγκεκριμένη αποστολή, είναι ανεξάρτητο. Νομίζω ότι έχει αρμοδιότητες Δεν νομίζω ότι οι πολίτες μας ε, είναι, ε, παρακολουθούν με χαρά τις ε, συγκρούσεις ανάμεσα σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα, το κάθε ταμείο είναι ένας διαφορετικός οργανισμός και δεν πρέπει να βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ε, έχουμε πολλά ε, πρακτικά ερωτήματα από τους πολίτες, πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ταμεία καλύτερη, ε, πώς μπορούν να υποφεληθούν από τη δράση τους κλπ. Αλλά τέτοιου είδους προβλήματα, αλλά προβλήματα τεχνικής φύσεως δεν παίρνουμε από τους δικούς μας πολίτες. Συνεπώς, δεδομένου ότι ο τίτλος της έκθεσης είναι πολύ σαφής, δηλαδή αφορά το πώς ε, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ε, αποτελεσματικότητα με τη συνέργεια έτυπα και άλλων διαφορετικών ταμείων. Νομίζω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Κάποιες ε, τροπολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν υποβληθεί και από εμένα και από άλλους συναδέλφους του ΕΛΚ και άλλων πολιτικών ομάδων. Επαναλαμβάνω λοιπόν, συμφωνώ με την αντιπρόεδρό μας. Το, η συζήτηση δεν θα πρέπει να εστιαστεί στις, στους καυγάδες ανάμεσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να γίνει σαφής, καθαρή, διάφανη συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα ταμεία. Υποστηρίζω λοιπόν τις ε, τροπολογίες ε, που πιστεύω ότι μας ε, βοηθούν να προχωρήσουμε. Ο εισηγητής. Grazie. Σας ευχαριστώ με τη σύνταξη αυτών των λύσεων ε, θα ηρεμήσουν ε, οι συνάδελφοι που πήραν το λόγο, αλλά θα, θα προσπαθήσω να το κάνω και εγώ από τώρα πριν από τη σύνταξη αυτή. Ακούστε, δεν θα με εξηγήσετε Σρέντερ, που χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα τις τροπολογίες σας. Οι τροπολογίες σας, εντάξει, μπορούν να γίνουν δεκτές όλες. Γιατί μπαίνουν σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που, στο οποίο συμφωνήσαμε από το ξεκίνημα ήδη στην Επιτροπή μας. Υπάρχει μια ε, ένα κενό maximum και μετά υπάρχει και αυτονομία και το κάθε ταμείο έχει το στόχο, του, το σκοπό του. Έτσι. Και αυτό όσον αφορά την γενική τοποθέτηση και αυτό που πολλές τροπολογίες από το ΕΛΚ υποστήριξαν όχι την αλλαγή του πλαισίου, αλλά την ενίσχυση του ειδικού χαρακτήρα μέσω της διατήρησης αυτού που αποδείχτηκε τελικά ένα σαν σημαντικό εργαλείο. Εντάξει, θα μπορούσε να βελτιωθεί, σίγουρα όμως δεν χρειάζεται να εγκαταληφθεί. Έτσι, η κοινωνική συνοχή, η γεωγραφική παρόμοια θα πρέπει να συμβαδίζουν. Η πρόθεσή μου είναι τίποτα. Δεν θέλω να αλλάξω από αυτή την τοποθέτηση που μας ενώνει. Απλά και μόνο θα ήθελα να προβάλλω μία ανησυχία μου που μου δημιουργείται από λίγες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και αυτές. Και η ανησυχία αυτή γίνεται εντονότερη από τη συζήτηση που γίνεται σε άλλους χώρους του Κοινοβουλίου, όχι εδώ, όχι εδώ σε αυτήν την Επιτροπή. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ένα μέρος του Κοινοβουλίου μας θα ήθελε να, θα ήθελε να ξεπεραστεί το κοινωνικό ταμείο των γεγονότων και αυτά τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται στο κοινωνικό ταμείο να πάνε στα άλλα ταμεία. Εγώ λέω ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει και αυτό, αλλά είναι σίγουρα λάθος. Λάθος. Γι' αυτό ακριβώς τόνισα τον κίνδυνο. Όχι, γιατί ε, αναφέρεται αυτός ο κίνδυνος εδώ σε εμά, αλλά είναι περισσότερο στην περιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, ίσως ε, για προφανέστερο λόγο. Εμείς ασχολούμαστε κυρίως περισσότερο με κοινωνικά θέματα, γι' αυτό ακριβώς το προσέχουμε αυτό περισσότερο. Είμαστε περισσότερο συγκεντρωμένοι πάνω σε αυτό. Εκεί μιλάνε τι γίνεται περιφερειακά, γεωγραφικά, άρα λοιπόν οι ανησυχίες δικές τους είναι κάπως διαφορετικές από τις δικές μας. Θεωρώ όμως ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δώσουμε την πραγματική αξία και στα δύο, περιφερικά και κοινωνικά, στα πλαίσια τους, της συνοχής, αλλά να μην απορρίψουμε την αυτονομία και την ύπαρξη του κοινωνικού ταμείου και την δυνατότητα να δίνει προσφαιρικό δίλια. Και μετά όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε βέβαια και στα διάφορα θέματα, τα δείτε και στις τροπολογίες και ε, θα τα συζητήσω και μαζί σας. Ευχαριστώ. η Πρόεδρος. Ε, εμείς αυτή τη γνωμοδότηση θα την εξετάσουμε την 1η Φεβρουαρίου και η Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων ε, θα το κάνει μετά στις 28. 27 σημείο τώρα της ημερήσιας διάταξης. Εκεί πάμε. Το λόγο έχει η κυρία Ομιν για τις τροπολογίες της, τις συμβιβαστικές για την πράσινη βίβλο, για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή συνταξιοδοτικά συστήματα. Κυρία Συγγήτρια, έχει τον λόγο. Collega's, mevrouw de voorzitter. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, σας έχω δώσει αντίγραφα του σχεδίου συμβιβαστικών τροπολογιών για το θέμα το οποίο συζητάμε τώρα. Αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες είναι ευθυγραμμισμένες ε, με αυτό το οποίο θεωρούμε και εγώ και οι πιο ως ε, βασικά σημεία αυτού του κειμένου. Θα σας πω ποιες είναι οι δύο παράγραφοι που χρειάζονται πιο λεπτομερή εξέταση. Λοιπόν, αρχίζω να μιλάω αγγλικά τώρα. Καταρχήν, διάβασα τις 460 τροπολογίες. Αν προσπαθήσει κανείς να κάνει τις συνήθεις συμβιβαστικές τροπολογίες, θα έπρεπε να τις βάλουμε στη σειρά, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε νέο κείμενο. Όμως κάτι τέτοιο θα μας έδινε μια μακροσκελέστατη έκθεση και δεν θα μπορούσε και να τη διαβάσει κανείς. Όλοι θέλουμε να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορούμε να δώσουμε την επόμενη εβδομάδα αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα, γιατί πρέπει η Επιτροπή να το λάβει υπόψη της το Φεβρουάριο και γι' αυτό προσπαθούμε να δώσουμε αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα. Πήρα λοιπόν τις ιδέες των συναδέλφων και τις έβαλα στην έκθεση. Αν επίσης δω, παραδείγματο χάρη, ότι η κυρία Φιγκερέιντο προτείνει μια τροπολογία ή ένα εναλλακτικό κείμενο και βλέπω ότι δεν συμφωνεί η πλειοψηφία για αυτό το νέο κείμενο, θα ζητήσω από την κυρία Φιγκερέιντο να το αποσύρει. Ή αν δεν το αποσύρει η κυρία Φιγκερέιντο, θα χρειαστεί να ψηφίσουμε. Με αρνητική πρόταση ψήφου από πλευρά τη εισηγήτρια, από δικιά μου πλευρά δηλαδή. Δηλαδή, τι προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ να δω τις ιδέες των συναδέλφων, να δω αν υπάρχει πλειοψηφία για τι ιδέε αυτέ, ούτω ώστε να τα συνδυάσω όλα αυτά. Δεν είναι μητρική μου γλώσσα τα αγγλικά. Και σας παρακαλώ να μου το πείτε αν υπάρχουν κάποιες διορθώσεις απαραίτητες, αν υπάρχει κάποια καλύτερη διατύπωση που έχετε να προτείνετε, παρακαλώ να μου το επισημάνετε για την αγγλική διατύπωση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας περιγράψω τώρα όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες, γιατί τα έχετε και μπορείτε να τα διαβάσετε. Καλύτερα να δώσω περισσότερο χρόνο στους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Και έχοντας ακούσει τα σχόλια των συναδέλφων, να απαντήσω εγώ. Γι' αυτό νομίζω καλύτερα είναι να σας δώσω εσάς το λόγο. Έχω τη συμβαστική τροπολογία 5 και τη συμβαστική τροπολογία 31 για τις οποίες υπάρχουν ακόμη σχετικές συζητήσεις και αύριο το πρωί θα προσπαθήσω να μιλήσω και με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να δούμε αν όντως το κείμενο στο οποίο καταλήξαμε είναι το σωστό. Και ανάλογα και με τις δικές τους αντιδράσεις θα σας προτείνω ένα νέο κείμενο ή θα το αφήσω ως έχει. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω εισαγωγικά και ελπίζω ότι θα καταλάβετε ότι δεν προσπάθησα να τα συμπεριλάβω όλα. Όλες τις ιδέες σας όμως προσπάθησα να τις ενσωματώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Όπως είπατε, θέλω και εγώ να επαναλάβω ότι έχουν γραπτό στις συμβαστικές σας προτάσεις οι συνάδελφοι. Παρακαλώ τη γραμματεία και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να στείλει στους συναδέλφους το κείμενο αυτό, γιατί διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσουν οι συνάδελφοι. Είπατε ότι όλοι είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν τις συμβαστικές αυτές τροπολογίες. Δυστυχώς όμως αυτοί που δεν είναι σκιώδεις εισηγητές ε, δεν έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν όλες τις τροπολογίες. Πολλοί από εμά ανακαλύπτουμε τώρα τις συμβαστικές προτάσεις τρο, τροπολογίες. Κυρία Όμεν Ρόιτεν, θα σας δώσω το λόγο στο τέλος. Ναι, μετά την παρατήρηση που κάνατε ήθελα να λάβω το λόγο τώρα. Είναι φυσιολογικό να συζητάμε τις τροπολογίες και μετά τη συζήτηση ο εισηγητής μαζί με τους κοιόδης εισηγητές θα κάνει τις συμβαστικές τροπολογίες. Και ήδη έχουμε, μία, έχουμε κερδίσει μια εβδομάδα. Είναι όμως απαραίτητο για να είναι ξεκάθαρο για τους συναδέλφους. Εγώ θα τα στείλω, όχι γραμματεία. Εγώ θα στείλω τις συμβαστικές τροπολογίες τη στιγμή που θα είναι έτοιμες. Για να μην υπάρξει σύγχυση. Αν τυχόν κάποιο κείμενο δεν ισχύει πλέον. Πρόεδρος, κυρία εισηγήτρια, ως πρόεδρος της Επιτροπής εγώ πρέπει να διασφαλίσω τις σωστές συνθήκες εργασίας για όλα τα μέλη της Επιτροπής. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση σήμερα. Νομίζω όμως ότι στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης καλό θα ήταν να μπορούν όλοι οι βουλευτές να έχουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις προτάσεις συμβιβαστικών τροπολογιών για ένα πολύ απλό λόγο. Να μπορεί ο κάθε συνάδελφος να εξετάσει υπό ποιες προϋποθέσεις αποσύρει την τροπολογία του. θα πρέπει οι συνάδελφοι που ενδεχομένω θέλουν να αποσύρουν την τροπολογία τους να δουν όλες τις συμβαστικέ τροπολογίε. Θα δώσω τώρα το λόγο σε αυτούς που ζήτησαν το λόγο, στον κύριο Όρη και στην κυρία Χάκιν. Αλλά α μην δώσουμε στα διαδικαστικά θέματα όλο μας το χρόνο, α ασχοληθούμε με το περιεχόμενο του κειμένου. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Ο κύριος Όρη και η κυρία Χάκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σωστό ότι η διαδικασία ε, δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όμως ε, θα συμφωνήσω με την Ρία. Είναι δύσκολοι οι συμβιβασμοί όταν έχουν υποβληθεί 460 ή 480 τροπολογίες. Και μάλιστα όχι σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές. Είναι δύσκολο η να έρθει σε επαφή με όλους τους συναδέλφους. Ε, ο χρόνος πιέζει. Δεν θέλουμε ε, να υπερβούμε τις προθεσμίες της διαβούλευσης. Ας ε, μην κατηγορούμε τη Ρία, ας κατηγορούμε τον εαυτό μας, κατηγορούμε τον εαυτό μας ή την υπηρεσία μετάφρασης που έπρεπε να βιαστεί πιο πολύ. Ε, μετά μπορούμε να μιλάμε για συμβασμούς ε, αν αυτοί βασίζονται σε μια συμφωνία. Ένα μεγάλο τμήμα του, κύματο, του κειμένου συγγνώμη, που έχουν μπροστά μας χρειάστηκε να τροποποιηθεί μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Οι τροπολογίε είναι πάρα πολλές. Ακόμα και στο εσωτερικό της ομάδας μας ε, δεν φαίνεται να συμφωνούμε πλήρως τα πάντα. Ε, εγώ δέχομαι το, τις συμβαστικές προτάσεις ε, και είμαι πρόθυμος να αποσύρω τις δικές μου τροπολογίες. Αν αρχίσουμε να ψηφίζουμε για 480 τροπολογίες, είναι προφανές κανένας δεν έχει διαβάσει όλες θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε ε, χωρίς να ξέρουμε τι ψηφίζουμε και θα χρειάζεται κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας να δίνονται εξηγήσει, οπότε θα κρατήσει εβδομάδες η ψηφοφορία. Νομίζω ότι υπάρχουν σημεία σύγκλησης, υπάρχει κοινός παρανομαστής, ε, παρόλο ότι υπάρχουν και σημεία διαφωνίας, ακόμα και στο εσωτερικό της κάθε ομάδας. Χαίρομαι που καταφέραμε να καταλήξουμε στο θέμα της ορολογίας τουλάχιστον. Γιατί όταν μιλάμε για το δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα, ε, αυτοί οι πυλώνες είναι κάτι διαφορετικό σε διαφορετικές χώρες. Χρειάστηκε να λύσουμε τέτοιου είδους προβλήματα, αρκετά τέτοιου είδους προβλήματα. οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν στην αναδιάρθρωση του πρώτου πυλώνα της αλληλεγγύης. Συμφώνησαν να πούμε ότι συμφώνησαν μάλλον ότι ε, οι απόψεις μας διαφέρουν σε ό,τι αφορά τους άλλους πυλώνες έτσι κι αλλιώ ε, δεν πρόκειται για κανένα διάταγμα, δεν πρόκειται για καμία απόφαση ή κάποια, κάποιο νομοθετικό κείμενο. Ε, είναι μια δημόσια διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου. Θα πρέπει να υποβάλουμε στην Κομισιόν τα σχόλιά μας για να τα συμπεριλάβει. Νομίζω ότι η μέθοδος που ακολουθούμε είναι η πιο ενδεδειγμένη. Και ως συντονιστή του ΕΛΚ νομίζω ότι με εξαίρεση ορισμένων ελάχιστων λεπτομεριών μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το συμβασμό και είμαστε πρόθυμοι να αποσύρουμε και ορισμένες τροπολογίες μας. Thank uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συγχαίρω την εισηγήτρια και χαίρομαι για τις ε, προσπάθειές της ε, το κείμενο να είναι συνεκτικό, λογικό και σαφές. Ε, διάβασα τις τροπολογίες επανειλημμένως και νομίζω ότι η εισηγήτρια έχει λάβει υπόψη πολλές, όχι όλες τις ιδέες, πολλές από τις ιδέες, τις βασικές. Και τις χρησιμοποίησε στο κείμενο, συμβαστικό της κείμενο. Χαίρομαι που αναφέρεται μόνο μία φορά σε κάθε θέμα, εκτός της αρχής επικουρικότητας, στο, στην οποία αναφέρεται δύο φορές. Ε, η υγεία και η ασφάλεια, για παράδειγμα, αναφέρεται μία φορά και πολλά άλλα ζητήματα στις τροπολογίες αναφέρονται μία φορά. Ε, θα ήθελα όμως διαμερικές διευκρινήσεις. Πρώτον, στον 8ο συμβασμό, στην 8η πρόταση συμβασμού, Μιλάει για την συμπερίληψη της μετρικής άδειας και της φροντίδας των ηλικιωμένων ε, ως ε, κανονική εργασία ε, σε ό,τι αφορά θέματα συνταξιοδότησης. Μια διευκρίνηση θα ήθελα τι ακριβώς εννοεί. Στην ένατη συμβαστική πρόταση είναι η μόνη πρόταση ε, για την οποία αμφιβάλλω συνολικά. Λέει θετικά κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην, ε, ε, στον υπολογισμό των συντάξεων των γυναικών. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί θετικά κριτήρια, λέγοντα θετικά κριτήρια. Δεν καταλαβαίνω πώ θα μπορούσαν να βρεθούν τέτοιου κριτήρια. Καταλαβαίνω το πρόβλημα βέβαια. Να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανεξαρτησία των πιο ηλικιωμένων γυναικών. Νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Μετά, στην 16η συμβαστική πρόταση, έχουμε ένα θέμα, δευτερεύον θέμα αρμοδιοτήτων. Ε, λέει να ενθαρρύνουμε την εργασία ε, πιο ηλικιωμένων ατόμων μέσω φοροαπαλλαγών ε, και φορολογικών κινήτρων. Δεν ξέρω αν έχουμε αρμοδιότητα για τέτοιο πράγμα. Στον συμβασμό 24 Ε, topical-based occupational pension systems, λέει το κείμενο. Τι σημαίνει αυτό? Θα ήθελα διευκρίνηση. Αυτά είναι βασικά τα σχόλιά μου και ερωτήσεις μου προς την εισηγήτρια. Ίσως μια-δυο άλλες ιδέες, οποίες δεν συμπερίλαβε, συμφωνώ με τον κύριο λέει ότι είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, αλλά ε, παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ε, για τις τροπολογίες 341 και 348 να ζητήσω από τον κύριο Τόμας Μαν διευκρινήσεις τι ακριβώς εννοεί. Νομίζω ότι την 341 την κατάλαβα, την 348 δεν είμαι σίγουρη ότι την κατάλαβα. Διευκρινήσεις λοιπόν από τον κύριο Τόμας Μαν. Υπάρχουν μια-δυο άλλες καλές ιδέες όπως σας είπα. Μία από αυτές την είπα την ανέφερα και προηγουμένω όταν μιλούσαμε με την Ουγγρική Προεδρία, υπάρχουν 40 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίε και πολλοί από αυτού ε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν ε, για τη βιωσιμότητα των συνταξιωτικών συστημάτων αν είχαν πρόσβαση στην εργασία. Ω ε, σκιώδη ηγετρία είμαι διατεθειμένη να αποσύρω τι δικέ μου τροπολογίε. Δεν έχω καταφέρει να μιλήσω με όλου μου του συναδέλφου αλλά νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα έχει γράψει η συγγετρία στο κείμενο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν νομίζω δικαιολογημένε οι ανησυχίε που εκφράσατε στην αρχή. Είναι δύσκολο να κάνουμε αυτή τη δουλειά με τόση πίεση χρόνου, αλλά αυτό αφορά και τις δύο επιτροπές, όχι μόνο την Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά και την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στην οποία επίσης είμαι μέλος. Κάναμε μία ψηφοφορία ε, σήμερα νωρίτερα και είδαμε ε, ότι ε, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εμπειρίες στα κράτη-μέλη και όλοι μας μεταφέρουμε την εμπειρία που έχουμε από το κράτος μέλος ο καθένας. Εδώ έχουμε 460 τροπολογίες και αυτό επίση οφείλεται στο ότι υπάρχει διαφορετική εμπειρία και τη διαφορετική μα εμπειρία προσπαθούμε να συνδυάσουμε σε μια κοινή έκθεση. Προσπαθούμε λοιπόν να εξομαλύνουμε το τοπίο και έχει σημασία το ότι κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλία ε, για μια πράσινη βίβλο. Υπάρχει το περιεχόμενο της ε, ε, πράσινης βίβλου και έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί φορείς και πολύ εντατικά με τα θέματα τα οποία πραγματεύεται η πράσινη βίβλο. Δεν ξέρω αν η εκδοχή που είχαμε τη Δευτέρα έχει τροποποιηθεί κατά πολύ ρία Πάντω θα μελετήσουμε τις ε, ε, συμβαστικέ τροπολογίε Στο χτεσινό κείμενο, στην πρώτη παράγραφο, εκεί που υποστηρίζεται η αρχή της επικουρικότητα και η συμβαστική τροπολογία 6, ε, για τα εξαιρετικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι κάτι που έχει προκύψει από την διαδικασία συζητήσεων με τους κοινωνικού εταίρους. Και στη συμβαστική λύση 7 με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Ακόμη συμφωνώ με την συμβαστική λύση 10 ε, δεν υπάρχει ενιαία ηλικία συνταξιοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Ε, πρόβλημα έχω με το θέμα που ανέφερε και η συγγήτρια σχετικά με τις ε, ε, ε, τροπολογίες πράσινη βίβλος και οι πυλώνες και εδώ είναι το 8ο ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα των κεφαλαιοποιητικών μοντέλων στις διευκρινήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία αγορά των συντάξεων λέγεται ότι η οδηγία αφορά τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα, άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα προς συζήτηση. Επίσης, ε, στις τροπολογίες της 22, 23 και 25, η ίδια η συγγήτρια αναφέρει το θέμα του δεύτερου πυλώνα και πάλι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν τροπολογίες και στο θέμα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Δεν συμφωνώ με τη χθεσινή εκδοχή που έχουμε ε, την συμβαστική τροπολογία για το 22 σχετικά με τα εμπόδια στην, κινητικότητα, στην εσωτερική κινητικότητα. Η εσωτερική κινητικότητα ε, είναι πολύ σημαντική για τα κράτη-μέλη και είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών Επίσης υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που δεν γνωρίζουν το θέμα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών, των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον ως ελάχιστη παροχή και ε, όταν μιλάμε για τις ελάχιστες παροχές θα πρέπει να δούμε και το αντίστοιχο κόστος. Και όταν υπάρχει ε, συμπληρωματικό κόστος για τα ιδρύματα επαγγελματικων ε, συνταξιδοτικων στεξιωτικών παροχών ε, υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που δεν έχουν καθόλου εμπειρία επί του θέματος. Και στο άρθρο 22 ε, αναγράφεται επίσης ότι θα πρέπει να διαγραφεί το τμήμα για τις χρονικές περιόδους και εδώ έχουμε το θέμα της φορητότητας των συντάξεων Στη Γερμανία υπάρχει μια διάταξη πενταετούς περίοδου. Στη Γερμανία έχουμε εμπειρία με τα επαγγελματικά ιδρύματα, ιδρύματα επαγγελματικών στεξιωτικών παροχών. Ε, υπάρχουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι συμφωνημένα από τους κοινωνικούς εταίρους και δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σαφώς υπάρχει διαφοροποίηση. Και μια τελευταία παρατήρηση. Σίγουρα υπάρχουν θέματα που μπορούν να συζητηθούν μόνο στην Οικονομική Επιτροπή ε, και άλλα θέματα είναι αρμοδιότητα μόνο τη Επιτροπή Απασχόληση. Αλλά υπάρχουν και θέματα που συζητούνται και στι δύο επιτροπέ και καλώ συζητούνται και στι δύο επιτροπέ και νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Σε γενικέ γραμμέ, λοιπόν, συμφωνώ με τι ε, συμβαστικέ τροπολογίε που διατύπωσε χθε η εισηγήτρια και πρέπει να δω τι σημερινέ συμβαστικέ τροπολογίε για να τι συγκρίνω. Υπάρχουν βέβαια πολλέ διαφορέ και θα δούμε αν θα υπάρξει αμφιλεγόμενη ψηφοφορία. Πάντως το ότι υπάρχει πολυμορφία πάντοτε είναι θετικό. Και ελπίζουμε από την πράσινη βίβλο να καταλήξουμε σε μια καλή λευκή βίβλο. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να βασιστούν στα θέματα αυτά τα οποία αναφέρονται στην ε, Πράσινη Βίβλο και να δίνουμε τα κατάλληλα μηνύματα προς τα κράτη-μέλη. Κύριος Κάσνερ, ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κοπίασε πολύ και κατέβαλε πολύ χρόνο για να έρθει σε επαφή όχι μόνο με τους χιώδης συγητές αλλά και με άλλους ενδιαφερόμενους συναδέλφους για να μπορέσει να καταλήξει σε αυτές τις συμβιβαστικέ λύσεις που μας έχει προτείνει. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να την ευχαριστήσουμε για το χρόνο και την προσπάθεια που κατέβαλε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι ε, σαφή και ευχαριστούμε πολύ τη Ρία για τα θέματα αυτά της ε, επικουρικότητας. Είναι ε, θέματα τα οποία τα έχει συμπεριλάβει και στις συμβιβαστικές τροπολογίες και πιστεύω ότι σωστά τονίζουμε την επικουρικότητα. Το ε, θέμα της δίκαιας αντιμετώπισης των γενεών επίσης είναι σημαντικό και θα πρέπει το διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, να τη συζητήσουμε και εδώ είχαμε την τροπολογία 138. Υπάρχουν, ε, υπάρχει πολυμορφία συνταξιδοτικών συστημάτων στην Ευρώπη και θα προσπαθήσουμε ε, να εξελίψουμε τις δυσκολίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε με το θέμα αυτό σε πολλές γενικές διευθύνσεις και κατέληξε στην Πράσινη Βίβλο μέσα από συζητήσεις σε πολλές γενικές διευθύνσεις και σε πολλές υπηρεσίες. Η δική σου έκθεση πρωτοβουλίας ξεκινά από την ε, Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει από την εμπειρία πολλών τομέων και πολλών ε, γενικών διευθύνσεων. Τα θέματα των κανόνων αφαιρεγγιότητας. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικά για μας την Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά θα πρέπει ε, να βρεθεί συμφωνία στην Ολομέλεια ε, του Κοινοβουλίου και όχι μόνο στη δική μας Επιτροπή. Υπάρχουν θέματα που αφορούν το δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα και θα μπορούσαμε εμείς να δώσουμε μια σωστή απάντηση με βάση τις δικές μας ιδέες από τη δική μας Επιτροπή. Τώρα, για άλλα συνταξιοδοτικά προγράμματα και για, για την φερεγγιότητα, για τη Solvency 2, ε, ξέρουμε ότι πολλές φορές απαιτούνται υψηλότερα επίπεδα και υψηλότερα αποθεματικά. Αλλά ε, επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, ε, θέλω να πω ότι μπορώ να συμφωνήσω με τις συμβιβαστικές τροπολογίες Ε, το έχουμε συζητήσει και στο ΕΛΚ και υπάρχουν κάποιες μικρές αποχρώσεις ε, που θα ήθελα να συζητήσουμε. Νομίζω ότι τα έχει συζητήσει και με άλλους σκιώδης συζητητές από άλλες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ άλλη μια φορά ε, και πιστεύω ότι καλά κάνουμε και προχωράμε γρήγορα γιατί το θέμα αυτό πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Thank you Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Είναι πολύ επικοδομητική η προσέγγιση της. Ε, καλά έκανε και αναδιέταξε. Την ε, γνωμοδότηση είναι, πιο, είναι πια σαφής, παρόλο οι πολιτικές μας πολλές φορές δεν είναι σαφείς. Ε, υπήρχαν πολλές ε, τροπολογίες κατά, ε, κατά των διακρίσεων ε, και της πρόσβασης κλπ. Ε, τώρα πια είναι πολύ σαφές το κείμενο. Το σημαντικό είναι ο πρώτος πυλώνας ε, να έχει ε, προτεραιότητα, το οποίο σημαίνει ότι οι συντάξεις θα πρέπει να ξεπερνούν το επίπεδο της Τα συστήματά μας πρέπει να λειτουργήσουν για τις γυναίκες, για τώρα τα ευάλωτα κομμάτια του πληθυσμού και Ιδιαίτερα δεδομένου ότι αλλάζει το πανόραμα στην εργασία, είναι ρευστό. Η συμβαστική πρόταση 9 ιδιαίτερως είναι σημαντική γιατί πρέπει να δούμε πώς ζίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους σήμερα, στο μέλλον ε, θα αλλάζουν εργασία πιο συχνά γι' αυτό ε, είναι με, μεγάλη σημασία τα στοιχεία της μεταφοράς των συντάξεων κλπ. Είναι πολύ καλό που η, ε, η συγγήτρια έχει λάβει υπόψη τις προτάσεις μας. Τώρα, ε, περιμένω να δω ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ε, για παράδειγμα, συμβαστική πρόταση 5, το πώς οι συντάξεις, πώς θεωρούμε θα έπρεπε να ε, αντιμετωπίσουμε τις συντάξεις μέσω του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τροπολογία 3.14 υπάρχει μια καλή ιδέα εκεί. Μετά η 16η συμβαστική λύση μας δημιουργεί προβλήματα σε ένα-δυο σημεία. Ενδεχομένως βέβαια δεν θα δημιουργήσει την υπόλοιπη επιτροπή προβλήματα, αλλά σε εμά δημιουργεί. Γενικά υποστηρίζουμε την μεγάλη πλειοψηφία των προτάσεων τη ηγητρια υπαρχουν Υπάρχουν μια-δύο παράγραφοι που θα θέλαμε να συζητηθούν, θα το κάνουμε κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα για να ε, καταλήξουμε στην οριστική μα θέση να δούμε ποιε τροπολογίε μπορούμε να αποσύρουμε. Θα το κάνουμε ως ε, ομάδα, συνολικά, συλλογικά. Monsieur Serkas, puis Monsieur Darden. Σέρκας, κύριος Darden. Εν συντομία, ο εισηγητή μα, ο κ. εισηγητή μα, ο κ. Νταρντέν, θα πει ποια είναι η άποψη τη ομάδα μα. Ε, θα είμαι σύντομο λοιπόν. Ε, να αναγνωρίσω το ρόλο τη ε, κ. Όμεν Ρόιτεν που βρίσκεται δύο βήματα πριν να ολοκληρώσει το έργο της. Για να αποφύγουμε προβλήματα της τελευταίας στιγμής, να πω τα εξής. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν ε, συνεργάστηκε με τους πιο εισηγητές. Ε, είναι ο μόνος ε, τρόπος να αντιμετωπιστούν οι 460 τροπολογίες. Αλλά μην ξεχνάμε για τη δημοκρατία. Όσοι έχουν υποβάλει τροπολογίες έχουν δικαίωμα έγκαιρα να γνωρίζουν αν οι τροπολογίες τους έχουν ληφθεί υπόψη στις προτάσεις, συμβαστικές προτάσεις. Συμβαστικές προτάσεις είναι καρπός συνεργασίας της εισηγήτρας με τους πιο εισηγητές. Θα πρέπει όμως όσοι υπέβαλαν τροπολογίε να ξέρουν. Συνεπώ, θα ήταν κρίμα τελευταία στιγμή να δημιουργηθεί πρόβλημα ε, διαδικασία. Μπορεί να λυθεί πολύ εύκολα. Να τη ζητήσω αύριο το πρωί, όταν θα έχετε, κυρία Συγγήτρια, κείμενο, ε, στείλτε μας το μέσο email, αύριο μεθαύριο, έτσι ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι συμβασμοί. Να μην δουν τους συμβασμούς πέντε λεπτά πριν ψηφίσουμε. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ε, θα ικανοποιούσαμε και την ανησυχία της Προέδρου και τις, ε, ε, τις επιταγές της ανάγκης για αποτελεσματικότητα. Να μην σκοντάψουμε τελευταία στιγμή γιατί βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας και έχουμε προχωρήσει πολύ καλά. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur Ευχαριστώ κύριος Νταρντέν. Καταρχήν, θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της και για τη συνεργασία. Για τις προσπάθειές της να συμπεριλάβει στη συμβαστική της πρόταση μια μεγάλη πλειοψηφία των προτάσεων προκειμένου το κείμενο να είναι ε, και σαφές και συνεκτικό δεδομένου ότι ε, οι διάφορες χώρες έχουν διαφορετικές εμπειρίες, οι διάφορα μέλη έχουν διαφορετικές ευαισθησίες. Δεν ήταν εύκολο το έργο της. Ε, το μήνυμά μας πρέπει να είναι σαφές προς την Κομισιόν και νομίζω ότι αυτό κάνει το, και το κείμενο της εισηγήτριας. Επί της ουσίας τώρα. Με μια πρώτη ανάγνωση των συμβαστικών της προτάσεων νομίζω ότι έχουμε σύγκληση σε πολλά σημεία. Για παράδειγμα, θεμελιώδης ρόλος του πρώτου πυλώνα και το γεγονός ότι οι άλλοι δύο πυλώνες είναι συμπληρωματικοί έναν του πρώτου η ανάγκη επιτυχίας της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ε, και η σημασία ε, η απασχόληση είναι όσο πιο ψηλή γίνεται, όσο πιο μεγάλη γίνεται. Η αναγκαία ε, συμμετοχή, στην ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και στην διαχείριση των συνταξιδοτικών συστημάτων. Όλα αυτά είναι τμήματα, κομμάτια τα οποία τα βλέπω στο συμβασμό. Μετά υπάρχει το θέμα των ορίων συνταξιοδότησης, ε, η έννοια της επικορικότητας και η ανάγκη να αυξηθεί η ε, πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης. Ε, όλα αυτά είναι σημεία σύγκληση. Παρ' όλα αυτά απομένει πολλή δουλειά και λίγος χρόνος δουλειά σε θέματα τα οποία είναι επίμαχα ακόμα. Για παράδειγμα, σύμφωνο σταθερότητας παράγραφος 5 και λοιπά. Είναι θέματα στα οποία θα έπρεπε ακόμα να προσπαθήσουμε να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις που θα γίνουν δεκτά, δεκτές στο μέλλον από όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης να δούμε αν η διευκρίνηση για την μεταφορά συνταξιδοτικών δικαιωμάτων είναι επαρκής. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο μέλλον. Και πέραν αυτών των σημείων να δούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της έκθεσης των άλλων επιτροπών, ιδιαίτερως Επιτροπής ΕΚΟΝ, και πώς οι δικές τους γνωμοδοτήσεις θα επηρεάσουν τη δική μας. πώς ε, θα ληφθούν υπόψη χωρίς να ε, ε, ξυλώσουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει εμείς. Τέλος, νομίζω ότι είναι σημαντικό σύντομα, γρήγορα να τεθεί στη διάθεσή μας ένα τελικό κείμενο και ένα είδος καταλόγου ψηφοφορίας, voting list, με τις τροπολογίες που καλύφθηκαν, αυτές που δεν καλύφθηκαν. Εγώ προσωπικά, σε συνεργασία με τον συντονιστή μου, θα πρέπει να ενημερώσουμε την ομάδα μας. Έτσι ώστε να διαπιστώσουμε σε ποιο μέτρο που θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις συμβασμούς τελικού κειμένου ή και να αποσύρουμε ορισμένες μας προτάσεις. Χρειαζόμαστε όμως αυτό το, την τελική εκδοχή του προσχεδίου και την voting list. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να συνομιλήσουμε με τους διάφορους ε, συναδέλφους μας. Η κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σκιώδης εισηγητρία για την ΚΟΕ, αλλά το, συνα... το συζήτησα με τον συνάδελφο Τόμας Χένλι και έχουμε υποβάλει από κοινού πολλές τροπολογίες και η Ήλτα Φιγκερέιδο και ο Πατρίκα Ρή επίσης έχουν υποβάλει τροπολογίες Πρέπει λοιπόν πολύ σύντομα να δούμε κατά πόσο αντικατοπτρίζονται οι δικές μας τροπολογίες σε αυτές τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Πολύ γρήγορα, με μια πολύ γρήγορη ματιά, βλέπω ότι υπάρχουν πολλές διαφορές στον τρόπο αντιμετώπισης. Καταλαβαίνω η δέσμευση και την πολλή δουλειά που κατέβαλε ε, η συνάδελφο ο και ε, είναι δύσκολη δουλειά και δεν το παραγνωρίζουμε αυτό. Αλλά όπως και πριν επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις. με τους συναδέλφους που είναι παρόντες εδώ προσπάθησα να καταλήξουμε σε κάποια αρχική κοινή θέση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές απόψεων. Δεν θα υποβάλουμε μια εναλλακτική πρόταση τώρα. Θα το συζητήσουμε άλλη μια φορά με τους αρμόδιους ε, ε, συναδέλφους, Πατρίκ Ρί και την Φιγκερέιντο. Παραμένουμε πάντως στις τροπολογίες μας ε, και ενδεχομένως θα έχουμε μια εναλλακτική πρόταση. Ακούστε να κάνω μερικές παρατηρήσεις επί της ουσίας. Για την ε, σημαντική λύση 5 το είπε ο Νταρντέν ότι πολλά θα έπρεπε ακόμα να επανεξετάσουμε, να βελτιώσουμε γιατί η σημερινή σύνταξη συνδυάζεται, συμβαδίζει με αυτό που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις μεταρρυθμίσεις τα λοιπά στον αφορά τις συντάξεις σε σημεία που δεν συμμεριζόμαστε απόλυτα με την προσέγγιση αυτή δηλαδή. Τώρα για να δούμε το σύνολο των συμβαστικών λύσεων. Εντάξει, ε, πιστεύουμε τον σκιωδή συγητή μα, αλλά τρία-τέσσερα για αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία είπα. Παράγραφος 12. Εκεί υπερασπίζεται κανείς μια μεικτή λύση και οδηγεί στην άποψη ότι σχετικά με τις συντάξεις μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα θα ήταν η καλύτερη εγγύηση για το συνταξιοδοτικό σύστημα το προσαρμοσμένο κατάλληλα. Προχωρούμε από μια χώρα που έχουμε μια σημαντική κοινωνική κινητοποίηση για να πούν όχι σε αυτή τη λύση. Γι' αυτό ε, δυσκολεύομαι να πω ότι είναι η, η καλύτερη εγγύηση για ένα συνταξιδοτικό καλό σύστημα. Είμαι κατά της άποψης αυτής, της σύνταξης αυτής και ακόμα στη 12α στη συμβαστική λύση για να δω το μη το λατινικό. Εντάξει, τι να σας πω τώρα εδώ, στο τέλος της παραγράφου η συγγήτριά μας τι προτείνει η μέθοδος συντονισμού έτσι επιτρέπει τρόπους εναλλακτικού χρηματοδότησης από τον πρώτο πυλώνα και αναρωτιέμαι τελικά από πίσω τι κρύβεται, άγγελος ή διάβολος. Πίσω από αυτή τη διατύπωση και ακόμα τελευταία επί της ουσίας παρατήρηση, παράγραφος 25, Ε, σε τοξικά ταμεία και και εντάξει λέτε κάτι το δεσμευτικό, αλλά ίσως θα πρέπει να δούμε και κριτήρια λειτουργίας. σημερίζουμε την άποψη αυτή. Αλλά αυτό το security που λέει εκεί, τι είναι, ε, να είναι φερεγγιότητα, τι να είναι. Ίσως θα μπορούσε να υπάρξει μια καλύτερη λέξη από το ασφάλεια που είναι στο τέλος της παραγράφου. Πώς είπατε? Ναι, παράγραφος 25, σε αυτήν αναφέρομαι τελευταία γραμμή της παραγράφου 25. Το ίδιο και για την επένδυση θα πρέπει να θεωρηθεί μακροπρόθεσμη γιατί αυτό ε, να το κάνει αυτός για να εκμεταλλευτεί την κατάσταση βραχυπρόθεσμα δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος, έτσι. Αυτά λοιπόν ε, οι παρατηρήσει που ήθελα να κάνω και η συγγήτρια έχει το λόγο. Παρακαλώ να είναι σύντομη βέβαια. Καταλαβαίνω ότι η συζήτηση αυτή έχει σημασία μεγάλη αλλά υπάρχει ακόμα μια σημαντική συζήτηση και έχουμε και εκπροσώπου από τους κοινωνικούς εταίρου. Γι' αυτό λοιπόν ε, να μην εξαντλήσουμε τον χρόνο που έχουμε, να αφήσουμε στο τέλο του και κάτι. Θα κάνω ό,τι μπορώ, πρόεδρε αλλά νομίζω ότι και οι συνάδελφοι στο πλαίσιο μιας καλής συζήτησης πρέπει να λάβουν τις απαντήσεις. Θα ξεκινήσω τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι θέλω διαφάνεια στη διαδικασία. Όλοι το θέλουμε αυτό. Ε, ήδη έγιναν κάποιες παρατηρήσεις και γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι θέλω μόλις έχουμε το κείμενο, το συντομότερο δυνατόν, να δώσω ένα αντίγραφο. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό, Πρόεδρε. Μόλις είναι δυνατόν. Αν θεωρώ ότι αύριο το απόγευμα είναι δυνατόν να το κάνω, θα το κάνω αύριο το απόγευμα, το συντομότερο δυνατόν. Και θα το κανονίσω με τους συναδέλφους, γιατί έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ότι όλοι, θα πρέπει να έχει, όλοι πρέπει να έχουν τις συμβαστικές τροπολογίες για να μπορέσουν να αντιδράσουν. Όλοι θέλουμε να αποκατασταθεί η ειρήνη στις σχέσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό. Για τις παρατηρήσεις που έγιναν, ξεκινώ με την κυρία Χάρκιν. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όλους σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και οι σκιώδεις εισηγητές δούλεψαν επίσης πολύ εντατικά και ήταν πολύ καλή η συνεργασία μας, άρα και εγώ σας ευχαριστώ. Και στο εξής δεν θα ευχαριστήσω κανέναν άλλον, σας ευχαριστώ όλους από τώρα για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις της κυρίας Χάρκιν. Επικουρικότητα, ναι, το ανέφερα δύο φορές. Επίτηδες το έκανα. Μετά, για την παράγραφο H, ε, ρωτάτε τι είναι τα θετικά κριτήρια και στη δική μου την ομάδα την ίδια παρατήρηση μου έκαναν. Να σας πω, γιατί με την κυρία Edith Bauer αυτό συζητήσαμε. Αν πούμε gender specific, σας ικανοποιεί αυτή η λύση. Αν έχετε εσείς να προτείνετε κάποια άλλη λέξη, προτείνετε την. Για το 16 για να λύσω ένα πρόβλημα και του συναδέλφου Τσάμπα Όρη. Στο τέλος της πρότασης να πούμε ενθαρρύνουμε το, τη δουλειά όλων και ζητεί από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν προσαρμοσμένα συστήματα απασχόλησης για όλους και να ενθαρρύνουν τα μέτρα για τη συνταξιοδότηση. Ε, ίσως να γίνει σαφέστερο το κείμενο αν προσθέσουμε κάτι. Εσείς ρωτήσατε ε, για τα παραδείγματα που αναφέρονται ως fiscal και security. Νομίζω ότι έχουμε δει από κάποιες χώρες ότι όταν οι πολίτες ε, ε, ζουν περισσότερα χρόνια, υπάρχουν κάποια, κάποιες διατάξεις από τις οποίες εξαιρούνται. Μου το εξήγησε η Σάρη και μπορεί να σας το εξηγήσει για να το καταλάβετε και εσείς καλύτερα. Έκανα τη διάκριση για να κατανοήσουμε καλύτερα την ορολογία και επίσης θα ήθελα να κάνω μια διάκριση σε αυτό που ανέφερε ο Τόμας Μαν για τα κεφαλαιοποιητικά και τα διανεμητικά συστήματα. Αν δεν το έχω εξηγήσει επαρκώς, αύριο θα επανέλθουμε. Τώρα προς τον Τόμας Μαν Υποθέτω ότι από χτες ε, έχεις διαβάσει το καινούριο κείμενο. Δεν έχουν αλλάξει πολύ αυτά που είπαμε χτες. Ε, μπορείς να είσαι ήσυχο ότι είναι σχεδόν ίδια με τα προηγούμενα που διάβασες χτες. Για κάποιους παραγράφους πρέπει να συμφωνήσουμε. Ελπίζω ότι αύριο θα τα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. την παράγραφο, 1, την παράγραφο 31 και την παράγραφο 5 θα πρέπει να τις εξετάσουμε για να δούμε αν είναι οι σωστές. Και όταν θα έχουμε το κείμενο, το συντομότερο δυνατόν θα το στείλουμε στους συναδέλφους. Εγώ θα ήθελα να έχουμε τις ελάχιστες, τα ελάχιστα πρότυπα, είπε. Όχι, όχι, δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι θέλω να έχω τα ελάχιστα πρότυπα. Πουθενά δεν μιλάω εγώ για ελάχιστα πρότυπα στις συντάξεις. Πουθενά. Κάπου υπάρχει λοιπόν κάποια παρανόηση. Ίσως ε, από την ε, ε, μεταφορά από τα αγγλικά στα γερμανικά ή τα γερμανικά στα αγγλικά. Πάντως εγώ δεν μίλησα πουθενά για ελάχιστα πρότυπα. Μετά, όταν μιλάμε ε, για την φορητότητα, αυτό ε, πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο ενός κοινοβουλίου. όπου η φορητότητα εξετάζεται από τους συναδέλφους διαφορετικά. Νομίζω ότι η πλειοψηφία θέλει περισσότερη φορητότητα από ό,τι θέλεις εσύ. Πρόσεξα όμως εγώ ιδιαίτερα στι παραγράφους για τη φορητότητα, γιατί και σε αυτές τις παραγράφους δεν θα δεις πουθενά Για να δω. Κοίτα να δεις τι λέει. Λέω. Επομένως, θεωρεί ότι τα εμπόδια στην εσωτερική και διασυνοριακή κινητικότητα πρέπει να αρθούν και θέματα όπως η δυνατότητα μεταφοράς κλπ. κλπ. πρέπει να αντιμετωπιστούν έχοντας κατά νου τις συνέπειες στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Δηλαδή, ε, ξέρω τι πιστεύει η πλειοψηφία και προσπάθησα να το βάλω αυτό ούτως ώστε να ικανοποιηθεί εσύ. Δηλαδή, λέμε πρέπει να αντιμετωπιστούν έχοντας κατά νου τι συνέπειε στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Προσπάθησα να λάβω υπόψη και τη δική σου θέση. Μετά προς τον κύριο Σέρκας. Ναι, όντως ήταν δύσκολη η συζήτηση και συνεργάστηκαν όλοι οι συνάδελφοι πολύ καλά. Και νομίζω ότι με τη δήλωση που έκανα μπορούμε αύριο το απόγευμα να στείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Και εγώ θα το ήθελα προς τον κύριο Νταρντέν. Ναι, για την 5 και την 31. Θα το συζητήσουμε αύριο με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ίσως μπορεί ο Γιάννη να έρθει σε επαφή με τους ε, υπευθύνου. Θα το συζητήσουμε. Για τη φορητότητα ήδη απάντησα στον κύριο Μαν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν για τη φορητότητα με αυτό που προτείνω. Λίγο πιο γρήγορα, κυρία Όμεν Ρόιντεν, λέει η πρόεδρο. Ε, πέντε λεπτά, πρόεδρε. Ναι, αλλά έχουμε άλλο ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Και έχουμε προσκεκλημένου. Ναι, πρέπει να απαντήσω σε άλλου δύο-τρει συναδέλφου. Παρακαλώ. Αυτά λοιπόν για τη φορητότητα και η κυρία Στάινρουκ και ο κύριος Μαν και ο κύριος Κάσλερ ε, βρίσκονται στην πηγή των ε, λύσεων τις οποίες έδωσα και ελπίζω να γίνει αποδεκτή η πρότασή μου. Προς τον κύριο Κάσλερ για την αφαιρεγγιότητα. Με η αφαιρεγγιότητα δεν είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, λέει η Πρόεδρος αυτές τις τροπολογίες θεώρησα μη παραδεκτές. Δεν είναι παραδεκτές. Άρα θεωρείτε ότι δεν χρειάζεται να απαντήσετε στον κύριο Κάστιο. Συνεχίστε κυρία Ομιρόιτεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα συζητήσουμε την αφαιρεγγιότητα όταν θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Γιατί ξέρετε ότι εμείς είμαστε αρμόδιοι η αρμόδια επιτροπή και θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Αλλά συμφωνώ απολύτω με την γνώμη του κυρίου Κάσλερ. Προ την κυρία Λάμπερτ, Πρώτο πυλώνα, επάρκεια κλπ. Θα τα συζητήσουμε αύριο. Αλλαγή τύπων εργασία. Νομίζω ότι είστε ικανοποιημένοι με την, συμβαστική μου λύση. Προς την κυρία Τσίμερ, ναι, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αλλά ελπίζω ότι και η δική σου πολιτική ομάδα θα μπορέσει να συμφωνήσει με τη νέα πρόταση. Θα είμαι διαθέσιμη και αύριο, αν θέλετε, για να σας τα ε, εξηγήσω άλλη μια φορά, γιατί τα έχω προτείνει αυτά τα οποία έχω προτείνει για την επόμενη ερώτηση μίλησα για, την τροπολογία 5, για τη συμβαστική τροπολογία 5 και 31. Θα κάνουμε μια νέα συμβαστική πρόταση. Για την παράγραφο 12 κάνατε κάποιες παρατηρήσεις που προκύπτουν από τις τροπολογίες της σοσιαλιστικής ομάδας και η χρηματοδότηση του πρώτου πυλώνα με εναλλακτικέ μορφές βγαίνει από μια τροπολογία των σοσιαλιστών. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ίσως να βρούμε μια λύση στο συντονισμό. Εγώ πήρα τις τροπολογίες, πήρα τις καλές ιδέες μέσα από τις τροπολογίες και τις δούλεψα με τους σκιώδεις εισηγητές για να καταλήξουμε σε συμβιβαστική πρόταση που νομίζω ότι είναι σωστή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Τελειώσαμε λοιπόν με το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Θα διεξαχθεί η ψηφοφορία την 1η Φεβρουαρίου. Βέβαια, μέχρι τότε και με τη φροντίδα της εισηγητριάς μας και με τη βοήθεια της γραμματείας Όσο γίνεται πιο σύντομα, σε όλα τα μέλη θα δοθεί ένας κατάλογος. Υπενθυμίζω βέβαια τους κανόνες λειτουργίας εδώ. Έχουμε την ε, γραμματεία, τη διοίκηση ακριβώς για να γίνουν σεβαστά όλα αυτά και ο καθένας να μπορεί να ξέρει πως έχει κατάσταση για τις τροπολογίες που θα καλύπτονται από τις συμβαστικές λύσεις και αυτό είναι ευθύνη της γραμματείας, έτσι και στη σχέση των ε, όλων. Και έτσι και όσοι καταθέτουν αυτές τις τροπολογίες θα μπορούσαν να τις αποσύρουν ε, σαν δείγμα καλής θέλησης απέναντι σε βαστικές. Και όπως το υπενθύμησε πολύ σωστά η κυρία Τσίμερ, δεν υποχρεώνει κανέναν να διαδικασία να αποσύρει την τροπολογία του, εντάξει, αλλά βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση μεταξύ δύο προσεγγίσεων, εντάξει, δείγμα καλή θέληση αυτή τη στιγμή που έχουμε μια συμβαστική λύση, θα, καλό θα είναι να αποσυρθεί. Τελικά όμως αν δεν ε, υπερψηφιστεί η συμβαστική λύση, δεν θα έχουμε τίποτα σαν ε, εναλλακτική λύση. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει κάτι το απαραίτητο στη διαπραγμάτευση η απόσυρση των τροπολογιών. Κύριο Ντερόζα, συγγνώμη για αυτόν και όπως επίσης και συγγνώμη για τους προσκεκλημένους μας. Ε, ερχόμαστε στο σημείο 28, το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έχουμε το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Ε, ανταλλαγή απόψε με κοινωνικού εταίρου, συζητή ο κύριο Ντερόσα. Το λόγο έχει ο κύριο Ντερόσα για να κάνει μια εισαγωγή στο όλο θέμα μα. Δεν θα με ακρηγορήσω γιατί έχουμε ήδη χάσει 20 λεπτά. Δεν είχαμε που δεν είχαμε πολύ χρόνο, τώρα έχουμε ακόμη λιγότερο. Θέλω να δώσουμε το λόγο στους κοινωνικούς εταίρους και δεν θα με ακρηγορήσω εγώ. Η έκθεση αφορά το μέλλον των, κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντο, τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενθαρρύνουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινή ωφελία σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Δίνω το λόγο όμως στους προσκεκλημένους μας κατευθείαν. Σας ευχαριστώ. Το λόγο θα βάλει η κυρία Α, Λίλιαν Βολοζίνσκι E ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να περιορίσω την παρουσίασή μου. Έχουμε λίγο χρόνο. Ε, εκπροσωπούμε τους εργοδότε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλω να επιμείνω στο ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφελία. Τις χρειάζονται όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαρτώνται περισσότερο από αυτές τις υπηρεσίες και την αξιοπιστία τους από ό,τι εξαρτώνται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι κοινωνικές υπηρεσίες ε, γενικού ενδιαφέροντος κοινωνικής ωφέλειας παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη καθώς επίσης και στην συνοχή οικονομική, κοινωνική και εδαφική. Μπορώ να συνεχίσω. Ωραία. Ε, η ε, προσβασιμότητα, η αξιοπιστία και η καλή ποιότητα αυτών των υπηρεσιών ζητώ συγγνώμη. Ε, ζητώ συγγνώμη. ζητώ όσους θέλουν να, το, να συζητήσουν να βγουν εκτός εθούσης και να σεβαστούμε λίγο την ομιλήτρια παρακαλώ πολύ. Αν έχετε συζητήσει παρακαλώ μεταξύ σας μπορείτε να βγείτε έξω. Είναι να περιμένετε μέχρι το τέλος της συνεδρίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ψηλή ποιότητα, αποτελεσματικότητα, προσβασιμότητα, ε, μη διάκριση και χαμηλό κόστος ε, ε, είναι βασικές, ε, τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, θεωρούμε ότι η οργάνωση και η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφέλεια είναι εθνική αρμοδιότητα. Θα πρέπει να τι μεταχειριστούμε με τη βάση αρχική επικορικότητα και αναλογικότητα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα όμως πάντοτε με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των κανόνων κρατικών προμηθειών, του, της ε, νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων είναι επαρκές. Λαμβάνει υπόψη την οικονομική και μη οικονομική πτυχή των υπηρεσιών αυτών. Συνεπώς δεν θεωρούμε ότι χρειάζονται περαιτέρω νομικές πρωτοβουλίες, νομοθετικές πρωτοβουλίες για αυτές τις υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καλωσορίζουμε τον οδηγό προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς πρακτικά θα εφαρμόζεται το νομικό πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφελία. Κανένα τέτοιο οδηγό θα επιτρέψει τα κράτη-μέλη και τι περιφέρειε να παρέχουν τέτοιου είδου υπηρεσίε με τον πιο οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Σε ό,τι αφορά την ε, ποιότητα των ε, διατάξεων ε, των υπηρεσιών, η όλο και περισσότερο περιμένουν όλη υψηλή ποιότητα και διαφάνεια. Ε, και οι χρήστες αλλά και οι φορολογούμενοι μεταξύ αυτών και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ε, υπηρεσίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κρατική χρηματοδότηση και μάλιστα δεδομένου ότι περνούμε ε, περίοδο περικοπών είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε λογαριασμό ακόμα και για το τελευταίο ευρώ που ξοδεύουμε. Καλωσορίζουμε τη δουλειά του, της SPC για το εθελοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κοινωνικών υπηρεσιών θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε ένα κοινό παρανομαστή και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφέλεια. Οι περισσότερες δυσκολίες αυτών των ε, υπηρεσιών αφορούν την ποικιλία, ποικιλία ε, προσεγγίσεων και ποικιλία αντικειμένου συμπεριλαμβανομένου και του outsourcing, της εξωτερικής ανάθεσης των υπηρεσιών αυτών. Εμείς είμαστε υπέρ της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, διότι αυτές θα έδιναν καινοτόμες λύσεις και πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων των αναγκών του υγειονομικού συστήματος, γύρανση, ε, ανεργία κλπ. Τελειώντα να πω το εξή, ότι αυτέ οι υπηρεσίε έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, ιδιαίτερα ε, στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, Απασχόλησης, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην, ε, και στην βελτίωση της συμμετοχή και ενσωμάτωσης. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποκτήσουν το κατάλληλο ε, ρυθμιστικό πλαίσιο που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα αποφεύγει ε, τις ε, παραβάσεις του, το, του, των κανόνων ανταγωνισμού. Ε, είναι ιδιαίτερο σημαντικό να διατηρηθεί χρηματοδότηση μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών ιδιωτικού δημοσίου τομέα Δεδομένου ότι τα δημόσια οικονομικά δέχονται όλο και μεγαλύτερε ε, πιέσει, ενώ τα κοινωνικά προβλήματα όλο και οξύνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρεμπέκα Σμιθ από την Business Europe. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη γιατί δεν έχουμε χρόνο. Καταρχήν θέλω να πω ότι και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα οι εργοδότες αποδίδουν μεγάλη σημασία σε αυτά τα θέματα και πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και το κόστος ωφελίας. Μας ενδιαφέρει επίσης να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και να λάβουμε υπόψη μας ε, διάφορες ε, αλλαγές όπως είναι η δημογραφική αλλαγή. Η πρόσβαση στις ε, κοινωνικές υπηρεσίες επίσης παίζει σημαντικό ρόλο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας. Οι υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν πολλά και να συμπληρώσουν συστήματα όπως τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και μπορούν να βοηθήσουν και συγκεκριμένου τομεί απασχόληση. Είναι σημαντικό να συνδυάσουμε την προσβασιμότητα και την ποιότητα με την αποτελεσματικότητα για να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα, ιδίω σε περίοδο δημοσιονομικών δυσκολιών. Και εδώ ε, υπενθυμίζω και την προσβασιμότητα και την αποτελεσματικότητα που ήταν θέματα που υπάρχουν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης του Δεκεμβρίου και στις συστάσεις του Τρίτου Φόρουμ για τις υπηρεσίες ε, γενικού ενδιαφέροντος. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κρίση οδήγησε σε επιδείνωση των οικονομιών των κρατών μελών, σε αυξανόμενο χρέος και έλλειμμα. Και είναι μια μεγάλη πρόκληση τώρα λόγω της επιδείνωσης ε, των πολιτικών να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές για να μειωθεί το επίπεδο του χρέους. Ε, σιγά σιγά περνάμε σε ανάκαμψη την οποία θέλουμε να επιτείνουμε και γι' αυτό θέλουμε να παραμείνουν ε, υγιεί τα δημόσια οικονομικά θα συνεχίσουν να παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες αποτελεσματικά και βιώσιμα. Στρατηγικές εξόδου από την κρίση θα πρέπει ε, να συνδυαστούν με στρατηγικές που θα επικεντρώνονται στην, ε, ε, σε μεταρρυθμίσεις της οικονομίας. Τονίζουμε λοιπόν την έμφαση που δίνουν τα κράτη-μέλη στην εξυγίανση του προϋπολογισμού. Όπως ήδη αναφέρθηκε από, από τη συνάδελφο, θα πρέπει να γίνουν αποτελεσματικές και αποδοτικές ε, οι ε, δημόσιες πολιτικές, ιδίως όταν δεν έχουμε επαρκείς πόρους και γι' αυτό θέλουμε ε, να βελτιώσουμε τη συνεργασία και την εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν κάποια όρια στις δυνατότητες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη δημοσιονομική πειθαρχία και, αυτό πρέπει, και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις θέσεις των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να ορίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Τα ορίζουν στα κράτη-μέλη ε, οι εθνικές και περιφερειακές και τοπικές αρχές και είναι φυσιολογικό το να μην υπάρχει νομικός ορισμός των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφελία, όπως η οικονομικές υπηρεσίες ε, ε, γενικού ενδιαφέροντος και ε, από το τρίτο φόρουμ του Οκτωβρίου του 2010 προέκυψε ότι η εφαρμογή των κοινών κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Όχι οι κανόνες αυτοί καθ' αυτοί, αλλά η εφαρμογή τους. Πρέπει να είναι ευκρινείς οι κανόνες και να γίνεται σωστά η εφαρμογή τους. Χρειάζεται καθοδήγηση και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχει ένα ζήτημα για τις κοινωνικές υπηρεσίες και το αν είναι οικονομικού ή όχι χαρακτήρα. Αυτό θα πρέπει κατά περίπτωση να αποφασίζεται γιατί δεν είναι ξεκάθαρο από τον ένα τομέα στον άλλο εξαρτάται από το είδος των δραστηριοτήτων. Για τους λόγους αυτούς δεν πιστεύουμε ότι χρειάζονται περαιτέρω νομοθετικά μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και η σύσταση του φόρουμ σχετικά με τον προτερισμό των δραστηριοτήτων που πρέπει ε, να διεξαχθούν. Αυτά είναι αρμοδιότητε των κρατών μελών, κατά τη γνώμη μα. Ακόμη, υπενθυμίζω ότι στο, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης του Δεκεμβρίου τα κράτη-μέλη δεν προέβλεψαν νομοθετικά μέτρα για τον τομέα αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα ήδη υπάρχουν μέτρα στη διάθεσή μας στον τομέα αυτό. Οι κανόνες τη Ευρωπαϊκής Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζουν την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και θα είναι χρήσιμη μια σχετική αξιολόγηση. Ήδη υπάρχουν μηχανισμοί του οποίους υποστηρίζουμε, παραδείγματο χάρη την ε, υπηρεσία πληροφόρηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν και οι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για του κανόνε τη εσωτερική αγορά το Single Market Act, ε, η νομική πράξη για την εσωτερική αγορά, που επίσης προτείνει κάποιους περαιτέρω κανόνες το εθελοντικό πλαίσιο για τι κοινωνικέ υπηρεσίε κοινή ωφελία, στο οποίο ήδη αναφέρθηκε συνάδελφο, επίση υποστηρίζεται από την Business Europe, γιατί είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και τι δημόσιε αρχέ και θα παρέχει εθελοντικέ κατευθυντήριε γραμμέ. Πιστεύουμε ότι είναι σωστέ αυτέ οι προτάσει, προτείνονται κοινέ αξίε και θα μα βοηθήσει να έχουμε κοινή κατανόηση για τι κοινωνικέ υπηρεσίε ε, κοινή ωφελία και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Εντείνεται το μήνυμα ότι είναι πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε την προσβασιμότητα με την αποτελεσματικότητα και την εφικτότητα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, α, να σας πω, συνάδελφοι, για τη συμμετοχή είναι μόνο γυναίκες ε, που εκπροσωπούν τους κοινωνικούς εταίρους. Άρα λοιπόν θα εξασφαλίσουν την ποιότητα της συναντησής μας. Η κυρία Ολρίκε Νουχάζερ. για το ε. Για τη CEP. Εκ μέρους της CEP θα σας μιλήσω καταρχήν για το νομικό πλαίσιο. Το ερώτημα είναι ποιοι τομεί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κοινωνική νομοθεσία. Εμείς ε, διαφωνούμε με ε, η εισαγωγή νομοθεσία για άλλε κοινωνικέ υπηρεσίε κοινωνική ωφελία, διότι ε, αυτέ είναι πολύ διαφορετικέ και πολύ συγκεκριμένες. Κάθε μία θα χρειαζόταν διαφορετική μεταχείριση και η συνολική έννοια των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφελία μόλι τώρα ξεκινάει να αποτελεί αντικείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν, ε, δεν έχει σαφή Ε, όσοι υποστηρίζουμε ότι δεν πιστεύουμε πω ένα νομικό πλαίσιο που θα κάλυπτε όλε αυτέ τις υπηρεσίε θα ήταν το καλύτερο ε, μέσο. Όμω, πιστεύουμε ότι αν μιλούμε για νομική βάση θα πρέπει να μιλήσουμε για μια κοινή βάση με τα άρθρα 9, 14 και το πρωτόκολλο. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες δημοκρατικών προμηθειών και την αθεώρησή τους, υποστηρίζουμε ε, εναρκτικές λύσεις έναντι των κρατικών προμηθειών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, ο, ιδιαιτέρως ε, επιτρέποντας ε, στις διάφορες αναλεκτικές δυνατότητες να λάβουν υπόψη τις καινοτομίες. Ε, υποστηρίζουμε επίσης την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης των κρατικών προμηθειών, διευκρινίζοντας την, ε, πιο, την έννοια της πιο οικονομικής προσφοράς, χω, προσφοράς, χωρίς να πρέπει να επιλέγουμε πάντοτε την πιο χαμηλή προσφορά. Διαφωνούμε με την νομοθεσία ε, σε κόρηση παροχής υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο, διότι δεν βλέπουμε την πρόσθετη αξία αυτής της νομοθεσίας. Αντιθέτως όμως, οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας ε, οι εξουσίε για αυτές τις υπηρεσίε ε, δίνουν τη δυνατότητα στι κρατικέ ε, αρχές με βάση τη Λισαβόνας να αποφασίσουν ποιε από τις γενικότερα από τις κοινωνικές υπηρεσίες θα θεωρήσουν υπηρεσίε κοινή ωφελία. Για την ρήτρα in-house υποστηρίζουμε την διαδημοτική συνεργασία και θέλουμε το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει μια πιο ευρεία προσέγγιση. Υποστηρίζουμε την ρήτρα in-house, ε, το υποστηρίξαμε και στον κανονισμο ε, ε, 3070 και θεωρούμε ότι θα πρέπει οι κανόνες εκεί των μεταφορών να εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες και όχι μόνο στις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά το κανονισμό, τους οριζόντους κανονισμούς με βάση το άρθρο 14 είμαστε υπέρ μιας προσέγγισης που θα συνδυάζει τον κανό, το θέμα με τον κλάδο, για παράδειγμα. Ε, όροι σε ό,τι αφορά θέματα κρατικών προμηθειών σε ρήτρε in-house θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για όλες, για όλες τις ε, δημόσιες κρατικές και όχι μόνο για τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, είμαστε υπέρ μια task force ψηλού επίπεδου με όλους τους ενδιαφερόμενους και είμαστε εναντίον της μείωσης του προπολογισμού, των προπολογισμού που υπάρχει για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, δημοσίων υπηρεσιών γενικότερα. Οι περικοπές που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μείωση των ελλημάτων πιστεύουμε ότι είναι ο λάθος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση των κρατικών υπηρεσιών, πιστεύουμε ότι η παροχή κρατικών υπηρεσιών είναι ένα από τα βασικά μελλοντικά προβλήματα των κοινωνιών μας. Το πόσο ο δημόσιος τομέας θα μπορούσε να συνεισφέρει στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών στο μέλλον είναι ένα από τα σημεία τα οποία θα πρέπει από κοινού να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρόλα Φίσπαρτ Πίτελ. European Federation uh, of Public Services κλπ. Έχετε το λόγο. Yes, thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων uh, Δημοσίων Ομοσπονδιών, η, ΕΠ, η EPSU, φορείς, ιδιαίτερα του δημοσίου τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα εκπροσωπούμεθα, στο μη κερδοσκοπικό τομέα και μερικές φορές ε, ε, και ε, στον τομέα όπου έχουμε κερδοφόρες επιχειρήσεις. Στη συζήτηση αυτή, αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να αναφέρω, στη συζήτηση αυτή για τις κοινωνικές υπηρεσίες, όπου μάλιστα η συνθήκη μας δίνει σαφώς εντολή δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η δουλειά που έγινε υπό Βελγική Προεδρία για την έγκριση του εθελοντικού πλαισίου ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Τώρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα οποία διαμόρφωσε η Βελγική Προεδρία και στην έκθεση γνωμοδότησης προς το σχέδιο έκθεσης ε, προς την ΙΜΚΟ, αυτό το οποίο αναγράφεται είναι ότι πρέπει να αναζητήσουμε πραγματιστικέ ρεαλιστικέ λύσεις. Η διάκριση μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών ε, δεν είναι χρήσιμη. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη βασική αποστολή των κοινωνικών υπηρεσιών και το ρόλο που έχουν στην κοινωνία μας και όχι το αν είναι οικονομικού ή όχι ενδιαφέροντος συμφωνώ με συναδέλφους από την πλευρά των εργοδοτών, όσο και αν σας εκπλήσει αυτό. Μόνο που τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι διαφορετικά. Πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγκαταλείψαμε κάπως την ιδέα ενός γενικού πλαισίου λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα και λόγω του ότι είναι δύσκολο να καθορίσουμε τι είναι κοινωνική υπηρεσία. Υπάρχουν πολλά είδη κοινωνικών υπηρεσιών όπως προέκυψε από τις συζητήσεις μας. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια πιο στοχευμένη προσέγγιση ανατομέα και αυτό το εθελοντικό πλαίσιο ποιότητας μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό σημείο σύγκρισης. Οι κοινωνικές υπηρεσίες χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο με τα χρήματα των φορολογουμένων και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε την ποιότητα, το δημοκρατικό έλεγχο και την λογοδοσία. Ένα επιχείρημα με το οποίο δεν συμφωνώ είναι ότι μέσω της εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν ξοδεύουμε δημόσια χρήματα. Αντιθέτως, οι εταιρικές σχέσεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα επίσης χρησιμοποιούν δημόσια χρήματα, χρήματα των φορολογουμένων, για να πληρώσουμε για τις ε, εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και οι δαπάνες αυτές και οι εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μακροπρόθεσμα είναι πιο δαπανηρές για τους ε, φορολογουμένους και όχι το αντίθετο. Και γι' αυτό κατά τη γνώμη μας δεν είναι η ε, πλέον σκόπιμη λύση. Λοιπόν, να δούμε μια ρεαλιστική προσέγγιση, να δούμε τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, να έχουμε σωστά σημεία σύγκρισης και πιστεύω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο ποιότητας για να δρομολογήσουμε πιλωτικά προγράμματα για την περίθαλψη των ηλικιωμένων, παραδείγματο χάρη. Η ποιότητα είναι η λέξη κλειδί για μας και αυτό το τονίζω ιδίως γιατί είναι μια αγορά εργασίας στην οποία υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες όπως γνωρίζετε και οι συνθήκες εργασίας ε, πολλές φορές δεν είναι καθόλου καλές και υπάρχει και υψηλό, υψηλός βαθμός εκμετάλλευσης. Η ποιότητα, το, η ποιότητα των υπηρεσιών λοιπόν συνδέεται και με την ποιότητα εργασίας και θέλουμε να υπάρχει υψηλός επαγγελματισμός στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει προστιθέμενη αξία από το να προσδιορίσουμε ένα καθεστώς γενικού ενδιαφέροντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών υπάρχει μεγάλη ποικιλία αυτών που παρέχουν υπηρεσίες και όλοι αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν κάποιες απαιτήσει ε, γενικών ε, υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και αυτά έχουν σχέση και με το δημοκρατικό έλεγχο και με την ε, λογοδοσία. Και εδώ αυτό που διαμόρφωσε η Βελγική Προεδρία είναι πολύ χρήσιμο. Ακόμη στην νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις Υπάρχουν θέματα που αφορούν ε, τις ε, ενδοϊπηρεσιακές υπηρεσίες, αυτήν την έννοια του in-house. Υπάρχουν οι συστάσεις για την ε, φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με τους στόχους της Βαρκελόνης και παρόμοια προγράμματα δράσης μπορούν να αναπτυχθούν ε, για την ε, μακροπρόθεσμη περίθαλψη ε, των ηλικιωμένων, των ψυχικά ασθενών, κατατίθεται δηλαδή μια πιο στοχευμένη προσέγγιση. Τις παρατηρήσεις μας τις έχουμε συμπεριλάβει σε ένα έγγραφο το οποίο υπάρχει διαθέσιμο από 18 συστάσεις έχουμε κάνει και κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις και ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο αυτό το έγγραφο. Σας ευχαριστούμε. Λόρα Τζόνς, τελευταία που λαμβάνει το λόγο αντιπρόεδρος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι αντιπρόεδρος της ε, ομάδας ε, υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος ε, της, ε, της Social Platform που είναι η μεγαλύτερη κοινωνική συμμαχία για την ε, κοινωνική δικαιοσύνη και τη συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρώπη με 42 ευρωπαϊκά δίκτυα μη κυβερνητικών ανώσεων και με πολλούς ενδιαφερόμενους, ε, πολλούς άλλους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τα τρία βασικά ζητήματα τα οποία μας προτείνατε. Να ξεκινήσω ε, για, με το νομικό πλαίσιο έχουμε τέσσερις λέξεις κλειδιά, καθολικότητα, εξειδίκευση, ευελιξία και αξιοπιστία. Σε ό,τι αφορά την καθολικότητα, να υπογραμμίσουμε ότι οι κοινωνικέ υπηρεσίε ε, κοινή ωφελία θα πρέπει να είναι διαθέσιμε και προσβάσιμε από όλου και όχι μόνο από του πιο ευάλωτου. Σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση, οποιοδήποτε νομικό πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ειδίκευση, την ειδικότητα, την, τον ειδικό χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών. Σε ό,τι αφορά την ευελιξία θα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και την, ε, ε και την ε, ε, κατακύρωση των, ε, της παροχής υπηρεσιών και να μην έχουμε μόνο τους κανόνες των κρατικών προμηθειών. Σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία χρειαζόμαστε ε, διευκρίνηση των κανόνων. Θα πρέπει οι κανόνες να είναι σαφείς, πιο σαφείς και προτείνουμε η Κομισιόν να δημοσιεύσει ένα, μια ανακοίνωση διερμηνευτική επεξηγηματική ενδεχομένω θα βασίζεται στον οδηγό που προετοιμάζει. Ε, έχει γίνει διαβούλευση για τι κρατικέ ενισχύσει, θα γίνει μια για τι κρατικέ προμήθειε και θα πρέπει οι υπάρχοντες κανόνες ε, να εξειδικευθούν με βάση τα απορίσματα αυτών. Τόσο ό,τι αφορά την βελτίωση ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Έχουμε την ποιότητα στη διαχείριση, την ποιότητα στην αγορά και την ε, ποιότητα στην ενίσχυση τη Ε, Σε ό,τι αφορά την πρώτη, Έχουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας ως ελάχιστο σημείο αναφοράς για τα κράτη-μέλη. Θα βελτιώσει την ε, κατανόηση της σημασία των υπηρεσιών αυτών στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, όπως σας είπα, ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των υπαρχόντων πλαισίων ή για την εκπόνηση νέων πλαισίων ε, τα οποία ε, θα παρέχουν την λεπτομέρειες για το πώς θα παρέχονται και θα αξιολογούνται οι υπηρεσίες. Ε, σε ό,τι αφορά την αγορά, την ποιότητα στην αγορά, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η πιο οικονομικά ε, χρήσιμη ε, πλεονεκτική πρόταση, προσφορά, όχι λιγό, η πιο οικονομική απλώς και επίση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ε, υποχρεωτικά συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητα και αρχέ ποιότητα. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα στην συμμετοχή, ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε την συμμετοχή των ενδιαφερομένων ε, και οι υπηρεσίες να είναι πιο εξειδικευμένε, πιο εξατομικευμένες. Τέλος, ο, λόγος ρόλος των υπηρεσιών αυτών στην κρίση ο κοινωνικό αντίκτυπος της ε, κρίσης ε, καθιστά όλο και πιο σημαντικές αυτές οι υπηρεσίε και συνεπώς ε, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί και ο προπολογισμό τους. Εδώ έχουμε τρία θέματα. Οι κοινωνικέ δαπάνε είναι επένδυση, είναι σημαντικές για την κοινωνική συμμετοχή, για την κοινωνική συμπερίληψη και είναι συμμετοχές αυτές τις υπηρεσίες και για την ολοκλήρωση της ε, αγοράς εργασίας. Καταρχήν, ε, να εστιαστώ στο πρώτο από αυτά τα θέματα. Οι κοινωνικές ε, δαπάνες είναι επένδυση γιατί επιτρέπουν στα, σε όλο τον πληθυσμό να συμμετάσχει στην κοινωνία και στην οικονομία. Και επίσης μειώνουν το κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης. δρούν επίσης πολύ προληπτικά και έτσι μας βοηθούν να αποφύγουμε πολύ πιο ακριβές θεραπείες αργότερα όταν ε, έχουμε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που αποκλείεται κοινωνικά. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική ε, συμπεριληψή θέλουμε ε, να μην αποκλείονται αυτοί που βρίσκονται στη πιο δυσχερή θέση. Σε ό,τι διάφορα αφορά την αγορά εργασίας μειώνεται η... με αυτές τις πλησίες βελτιώνεται το επίπεδο υγείας το οποίο σημαίνει ότι θα είναι πολύ καλό βέβαια αυτό για την αγορά εργασίας στο μέλλον. Ε, εδώ να υπογραμμίσουμε τη σημασία του κοινωνικού τομέα στην δημιουργία θέσεων εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τις πέντε σας. Ήταν κάτι το πολύ σημαντικό για μας, το ξεκίνημα της διαδικασίας ε, γύρω από τον εισηγητή Ρώσα, να σας ακούσαμε και τις πέντε σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας και για τα μέλη που είναι εδώ μαζί μας και θέλουν να παρακολουθήσουν ακριβώς προσεκτικά το θέμα μέχρι να πάει στην Ολομέλεια. Ήταν πολύ ωφέλιμο να ξεκινήσουν με τις παρεμβάσεις σας. Είστε οι πρώτες που συναντάμε για τη μελλοντική αυτή έκθεση του Ντερός. Δυστυχώς δεν είχαμε το χρόνο διάθεσή μας για να έχουμε και περισσότερη συζήτηση μαζί σας αλλά καλό ήταν που ήρθατε εδώ. Είσαστε το πρώτο φως που μας δόθηκε και που μας ε, προσκαλεί έτσι να συνεχίσουμε τη διαδικασία γύρω από την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τους διερμηνείς που μας συνόδευσαν σε αυτήν την παράταση ε, εδώ στο ξεκίνημα της χρονιάς. Και εντάξει, για την επόμενη συνάντηση, λοιπόν, 15-16 Μαρτίου, το θέμα του κ. Ντυρόσα. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε όλοι μέχρι το τέλος της συνάντησή μας και σας περιμένω δίπλα για ένα φιλικό ποτηράκι, για μια πρόποση ακριβώς για να ξεκινήσουμε καλά και θα έχουμε και υπό την προεδρία της κ. Λίν την επόμενη συνάντηση την 1η Φεβρουαρίου.